Αγαπητοί συνάδελφοι, αρχίζοντας αυτή τη συνεδρίαση της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να συγχωρήσετε τον Πρόεδρό μας, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορεί να παρευρεθεί και από τις 4 θα έχουμε τον συνάδελφο Μπάρστατ και Στάς ε, από τις 4 η ώρα ε, και στο ενδιάμεσο. Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι η ακρόαση του κυρίου την Βίρντε, Βίρντα με συγχωρείτε, πρώην μέλους του ελεγκτικού συνεδρίου που προβλεπόταν για τις 3 Μαρτίου αναβάλλεται για τις 17 Μαρτίου. Πρόκειται για μια ακρόαση που αποφασίστηκε από τους συντονιστές. Λάβατε την ημερήσια διάταξη τα πρακτικά μάλλον της τελευταίας συνεδρίασης, τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης. Υπάρχουν παρατηρήσεις σχετικά με τα πρακτικά αυτά. Όχι, θεωρώ συνεπώς ότι τα πρακτικά αυτά υιοθετούνται, εγκρίνονται και σας προτείνω να περάσουμε στην ψηφοφορία όπως σας ανακοινώθηκε προτείνω ε, να να, να ψηφίσουμε με τις ηλεκτρονικές κάρτες και όχι με ανάταση χειρός. Έχουμε μια πρώτη εισήγηση, Καταλήν Σορίν Ιβάν, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά πολέμηση απάτης, ετήσια έκθεση 2009. Παράγραφος, ο πρώτη παράγραφος, τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Le vote est ouvert. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Δεν λειτουργεί το δικό σας. Donc l'amendement est repoussé. Amendement numéro 5. Le vote est ouvert. Απορρίπτεται. Ε, τροπολογία 5. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Γίνεται αποδεκτή η τροπολογία. Τροπολογία 7. Αρχίζει η ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας. Γίνεται αποδεκτή η τροπολογία. Τροπολογία 8. Με ξεχωριστή ε, ψηφοφορία το πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε για το πρώτο τμήμα. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Μετά έχουμε μια προφορική τροπολογία για το δεύτερο τμήμα. Ποιος θα παρουσιάσει την προφορική τροπολογία. Κύριε Ανδρεάς, θα παρουσιάσετε την προφορική τροπολογία. η κυρία Ανδρέασεν. Κύριε Ανδρέασεν, η προφορική σας ε, τροπολογία. Έχετε στον ε, κατάλογο, στον κατάλογο ψηφοφορίας. ζητά από την Κομισιό να αναλάβει τις ευθύνες όσον αφορά την διασφάλιση της συμμόρφωσης των κρατών μελών προς τις υποχρεώσεις γνωστοποίηση έτσι ώστε να παρέχουν αξιόπιστα και συγκρίσιμα στοιχεία Ακόμη και αν αυτό απαιτείται, απαιτεί η Επιτροπή να καθιερώσει κάποιο σύστημα κυρώσεων για τη μη συμμόρφωση με τις εν λόγω υποχρεώσεις. Δεύτερο τμήμα λοιπόν της τροπολογίας 8 με την προφορική ε, τροπολογία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται τροπολογία 14, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται τροπολογία 15, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται Τροπολογία 16. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται τροπολογία 17 με μία προφορική τροπολογία. Ε, η κυρία Μάκοβέη. Ναι, η προφορική τροπολογία για ε, ε, να, αντικαταστήσουμε την Εστονία. Από την Ισπανία. Ο κύριος Γκάγια, Κύριε Πρόεδρε, η πολιτική μου ομάδα ε, έχει μια προφορική τροποποίηση να ζητήσει στην προφορική τροπολογία. Γιατί πιστεύουμε ότι δύο πολύ σημαντικές λέξεις λείπουν. Η διατύπωση της κυρίας Μακοβέη επιτρέπει την εξή ερμηνεία. Το ίμιση των χρημάτων, των ποσών δηλαδή, που έχουν πάει στις χώρες αυτές ε, ε, ήταν αντικείμενο απάτης ή θύμα απάτης. Ε, δεν είναι αυτό, δεν λέει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι οι μισές ατασταλίε, ανομαλίε, irregularities, ε, είναι λόγω απάτης. Και από αυτή την αλλαγή θα εξαρτηθεί και η υπερψήφιση της τροπολογίας από εμά. Να τα διαβάσω στα αγγλικά πώς θα έχει. Ανησυχεί για το ύψος ή το ποσό των απατών σε σχέση με τις ατασταλίες στους ιδίους πόρους για τα κράτη-μέλη Αυστρία, ε, Ισπανία, Ιταλία, Ρουμανία και Σλοβακία. Καθώς τα κρούσματα αυτά ε, απάτης είναι το μισό των ατασταλιών ε, στα ε, κράτη-μέλη. Καταλαβαίνετε τι λέω και θα εξαρτηθεί αν θα ψηφίσουμε την τροπολογία αυτή. Ναι, για μένα το κείμενο είναι σαφές, αλλά συμφωνώ με αυτή την προφορική τροπολογία. Καταλαβαίνω καλά ότι προσθέτουμε τις δύο προφορικές τροπολογίες Πολύ καλά. Λοιπόν, τροπολογία 17 με τις δύο προφορικές τροπολογίες. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορίες, Εγκρίθηκε. Τροπολογία 18. Αρχίζει η ψηφοφορία. Κύριε Γκαγιέρ. Η ομάδα μας έχει αντίστοιχο πρόβλημα. Δεν ξέρω, μπορεί να φταίει η, διερμηνία, η μετάφραση, συγγνώμη εδώ, η γραπτή μετάφραση, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να μας εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς καταλήγει σε αυτές τις εκτιμήσεις για τα ποσοστά απάτης και ατασταλιών. Εμείς δεν αμφισβητούμε τους αριθμούς, τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γι' αυτό προτείνουμε να πούμε. Ανησυχεί από ε, τις ύποπτα χαμηλές υποτιθέμενες περιπτώσεις απάτης κτλ. Yes. Η κυρία Μακοβέη, τι λέει, ο πρόεδρος. Στη 18 λοιπόν με αυτή την προφορική τροποποίηση ψηφίζουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Βοτικλού. Πέρα της ψηφοφορία. Δεν λειτουργεί το μηχάνημα. Δεν λειτουργήσε. Ξαναρχίζουμε την ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία ξανά. Πέρα της ψηφοφορία. εγκρίνεται. Τροπολογία 19 αποσύρεται κυρία Ανδρέασεν. Ναι. Αποσύρεται. Ναι. Μετά έχω μια προφορική τροπολογία του εισηγητή. Υπαριθμών ε, με β. Έχετε Ας ψηφίσουμε λοιπόν για αυτήν την προφορική τροπολογία εφόσον την έχετε στο φάκελό σας. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Τροπολογία 20. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας απορρίφθηκε. Συμβιβασμός Α. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 23 με μια ε, προφορική τροπολογία Δ που έχετε στο φάκελό σας. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας απορρίφθηκε. Τροπολογία 24. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Τροπολογία 25. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Τροπολογία 26 σε τρία μέρη. Πρώτο τμήμα, πρώτο μέρος, αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Δεύτερο τμήμα, αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τρίτο τμήμα, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίφθηκε. Τροπολογία 27 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίφθηκε. Τροπολογία 28 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας Απορρίφθηκε. Δεύτερο τμήμα αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 29 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Συμβιβασμός Β αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 32. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 33. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 34. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Προτείνω να ψηφίσουμε μαζί τις τροπολογίες 35-41. On block. Έχει κανείς αντίρρηση, όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν για όλες τις τροπολογίες από την 35 έως την 41. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίθηκε. Κυρία Μακοβέη. Για την προφορική τροπολογία για την 40 να διαγράψουμε τη λέξη presidency. Δεν ψηφίζουμε λοιπόν για αυτήν την πρόταση. Τη γραμματεία το σημειώνει αυτό. Τροπολογία 35. τροπολογία 1. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Αρχίζει η ψηφοφορία. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Ο συνάδελφος Γκάιερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς πιστεύουμε ότι εδώ υπάρχει ένα διαδικαστικό πρόβλημα. Διότι στην έκθεση αυτή, ε, πρόκειται για έκθεση πρωτοβουλίας, ξέρετε. Και η διαδικασία που προτείνει η κυρία Ανδρέα Σεν, κατά τη δική μας ανάγνωση, δεν είναι δυνατή. Και θα παρακαλούσαμε να απορρίψετε αυτή την τροπολογία, γιατί αυτό που επιδιώκει τώρα η κυρία Ανδρέα Σεν θα πρέπει να αποφασιστεί από τις πολιτικές ομάδες στη διάσκεψη των Προέδρων και όχι εδώ. Madame Κύριε Ανδρέασεν, νομίζω ότι αναφέρεται σε διαδικαστικό θέμα. Νομίζω ότι το θέμα αυτό, το θέμα εδώ είναι αν αυτό ψηφίζεται εδώ ε, στην Επιτροπή, αν θα πρέπει να ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Δεν έχω τίποτα να πω. Η γραμματεία μου λέει ότι ε, δεν είναι παραδεκτή ε, τροπολογία. Γιατί τότε μπήκε στον κατάλογο των ψηφοφοριών. Σας προτείνω λοιπόν να θεωρείται ως μη παραδεκτή την τροπολογία σύμφωνα με τις συμβουλές της Γραμματείας και βεβαίως ε, η συνάδελφος θα ξαναπαρουσιάσει την τροπολογία στην Ολομέλεια. Τροπολογία υπαριθμών 3. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τροπολογία 3. Τροπολογία 3. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Περνάω στην τελική ψηφοφορία όλη της γνωμοδότηση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε με 19 ψήφους υπέρ, δύο αποχές και καμία αντίθεση, καμία ψήφο κατά. Θα ήθελα κύριε Γκάιερ να συγχαρείτε τον εισηγητή για αυτή τη γνωμοδότηση εφόσον δεν είναι παρόν. Τώρα περνάμε στην έκθεση για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, γνωμοδότηση Παράγραφος 1. Η τροπολογία 1. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Le vote Υπέρασε. Εγκρίνεται. Η τροπολογία υπάρχουν δύο. Ψηφίζουμε, παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. τροπολογία υπαριθμών 3, άρχιδη ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Η 4 ψήφι υπέρ. Μάλλον άρχεται ψηφοφορία, συγγνώμη. Πέρασε. Απορρίπτεται. τροπολογία υπαριθμών 5, ε, άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Επτά αρχή ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 6. Αρχή ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 8. Αρχή ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται η τροπολογία παριθμών 9 άρχη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται η 10 άρχη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η τροπολογία παριθμών 11 άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η τροπολογία υπαριθμών 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η τροπολογία υπαριθμό 15 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η συμβιβαστική υπαριθμό 1 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και περνούμε στην τροπολογία 18 αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. Η 19, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η συμβαστική παριθμό 2, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και παίρνουμε στην οριστική ψηφοφορία. Τελική τώρα άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 19 ψήφοι υπέρ, 2 κατά και καμία αποχή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή που είναι υποφαινόμενος. Συνεχίζουμε. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη τώρα, ακολουθεί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 Παρνάμε Witam serdecznie w kolejnym punkcie naszego posiedzenia. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης, αγαπητοί συνάδελφοι, το σημείο είναι παριθμών 6. Απαλλαγή 2009, παρουσίαση των συστάσεων του Συμβουλίου από τον κύριο Σόλτ Μπέξεϊ, Υπουργό Εθνικής Οικονομίας της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας παρουσία του κυρίου Αλγκέρντα Σέμετα του Αρμοδίου Επιτρόπου για τη Φορολογία και Τελωνιακή Ένωση, τον έλεγχο και την καταπολέμηση τη απάτη, τον οποίο και καλώ ορίζω. Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο και ονόματο τη Ουγγρική Προεδρία. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι κύριοι και κυρίες ευρωβουλευτές, κύριε Πίτρο Σεμέτα. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω που ως εκπρόσωπος της Προεδρίας και πριν αρχίσω την ομιλία μου σας καλωσορίζω εδώ πριν από λιγότερο δύο χρόνια ήμουνα κι εγώ εδώ, ευρωβουλευτής. Έτσι τα φέρνει η ζωή όμως. Ελπίζω ότι με την παρουσία μου σήμερα από την πλευρά της ε, Προεδρίας να έχω μια ακόμα πιο στενή και αποδοτική σχέση στη συνεργασία μας. Μετά από αυτή την μικρή εισαγωγή Αρχίζω την ομιλία μου. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, είχα έναν κανόνα να μιλάω στη μητρική μου γλώσσα. Θα τον παραβώ όμω. Σήμερα θα μιλήσω στα αγγλικά, θα είναι πιο εύκολο έτσι για εσά να με παρακολουθήσετε. Με μεγάλη ικανοποίηση και τιμή έρχομαι να σας, στην Επιτροπή σας σήμερα, όπως προβλέπουν οι συνθήκες, για το ρόλο της Προεδρίας με βάση τη διαδικασία ετήσιας απαλλαγής και να σας και τα, τις θέσεις του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή για τον, την εκτέλεση μάλλον του προπολογισμού 2009 Κομισιόν. Αυτό εγκρίθηκε από το ΕΚΟΦΗΝ στις 15 Φεβρουαρίου και εστάλει στο Ευρωκοινοβούλιο η απαλλαγή μετά από μια εκτενή ανάλυση των τελευταίων μηνών όσον αφορά την εκτέλεση του Γενικού Προπολογισμού της Ένωσης για το Οικονομικό έτος 2009 ε, από την Επιτροπή με βάση και τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ετήσια έκθεσή του. Καταρχήν, ποια είναι τα τέσσερα βασικά σημεία που θα θέλω να τονίσει το Συμβούλιο στις συστάσεις του. Πρώτον, σημειώνουμε τις τι βελτιώσει που επισήμανε και το Εκδοτικό Συνέδριο, ιδιαίτερα στην ε, πολιτική συνοχής και στην μείωση του ποσοστού λάθους γενικά. Δεύτερο, το Συμβούλιο ωστόσο ανησυχεί διότι η γνώμη του Ελεκτικού Συνεδρίου δεν συμφωνεί με ένα σημαντικό κομμάτι του προϋπολογισμού και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να βελτιώσουν την περαιτέρω διαχείριση και σωστή εκτέλεση ε, δαπάνης των κοινωτικών κονδυλίων. Τρίτον, το Συμβούλιο θεωρεί ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο για την περίοδο προγραμματισμού είναι σωστό, αλλά περαιτέρω απλούστευση των προγραμμάτων και των συστημάτων είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται. Και τέσσερα, το Συμβουλίο επισημαίνει τη σημασία ε, διαφανών συστημάτων ανάκτησης κονδυλίων και οικονομικών διορθώσεων ε, εκ μέρους της Επιτροπής και στα κράτη-μέλη. Κυρίες μου και κύριοι, αγαπητοί πρώην συνάδελφοι, τώρα θα μπω σε λεπτομέρειες όσον αφορά τα σχόλια και τους λόγους που οδήγησαν το Συμβούλιο στη σύσταση απαλλαγής. Πρώτον, το Συμβούλιο σημαίνει με ικανοποίηση την δήλωση του συνεδρίου ότι για τρίτη φορά στη σειρά οι αιτήσιοι λογαριασμοί της Ένωσης παρουσιάζουν σωστά την οικονομική θέση της Ένωσης όσον αφορά τις διάφορες πράξεις και την ε, ταμιακή ροή. Το Ελληνικό Συνέδριο επίση θεωρεί θετικό την βελτίωση στη διαχείριση κονδυλίων όσον αφορά την νομιμότητα των πράξεων. Τα τελευταία χρόνια το ποσοστό σφάλματος συνεχώς μειώνεται. Τώρα περίπου υπολογίζεται αυτό γύρω στο μεταξύ 2 και 5%. Το Συμβούλιο είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένο λόγω των βελτιώσεων σε θέματα πολιτικής συνοχής, όπου ελήφθησαν σημαντικά μέτρα και από την Κομισιόν και από τις κυβερνήσεις και τώρα άρχισαν να αποδίδουν. Σημαντική μείωση των εκτιμόμενων δαπανών στον τομέα αυτό που δεν έχουν επιστραφεί με βάση ε, το συμβουλίο που έπεσαν από το 11% τα τρία προηγούμενα χρόνια στο 3% μείωση. Αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα για τους Ευρωπαίους πολίτες και φορολογούμενους. Γιατί τώρα που ζούμε την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, πολλές χώρες υποχρεωμένες να περικόπτουν τους προπολογισμούς τους, οι δαπάνες υπό αυστηρό έλεγχο, και εγώ ως Ούγγρος τα ξέρω πολύ καλά αυτά, οι πολίτες αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στο να δαπανώνται σωστά τα κοινοτικά κονδύλια. Οι βελτιώσεις λοιπόν που τις επισήμανε και τις ε, θεώρησε θετικές στο ελληνικό συνέδριο και όλοι μαζί σας ελπίσουμε ότι η προοπτική θα είναι θετική και εφ' εξής. Παρ' όλα αυτά τα θετικά μηνύματα όμως, το συνολικό αποτέλεσμα δεν είναι και πάρα πολύ ικανοποιητικό. Χρειάζεται σκληρή προσπάθεια να βελτιωθεί η κατάσταση ένα μεγάλο τμήμα πληρωμών από τον προπολογισμό επηρεάζονται ακόμα από σφάλματα. Συστήματα εποπτείας εν μέρη είναι αποτελεσματικά. Και αυτό αφορά πολλές πολιτικές. Γεωργία, φυσικούς πόρους, όπου το σφάλμα υπολογίζεται από το Ελληνικό Συνέδριο σε αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Το Ελληνικό Συνέδριο λοιπόν Πρέπει να αιτιολογήσει βέβαια τη γνώμη του για το 2009. Κύριος στόχος είναι να πετύχουμε μια θετική διασφάλιση, το λεγόμενο θετικό Αυτό δεν έχει επιτευχθεί. Συνεπώς το Συμβούλιο επισημαίνει τη σημασία του να βελτιωθεί αυτό το σύστημα εποπτείας των δαπανών και για τώρα και για τα επόμενα έτη. Και ένας καλός τρόπος να μειωθούν οι παρατυπίες για να έχουμε πιο καλά αποτελέσματα είναι ακριβώς αυτό. Αλλά αυτό μπορεί να τεθεί και ως ερώτημα. Το Συμβούλιο θεωρεί ότι οι βελτώσεις που επετέφθησαν αυτή τη χρονιά και η συνολική μείωση του ποσοστού σφάλματος σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο ρυθμιστικό πλαίσιο που ορίστηκε για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Ποιο σαφείς κανόνες, πιο αποτελεσματική εποπτεία. Προβλέπονται από τους νέους κανονισμούς το ποσοστό επιστροφών σε σχέση με τη νέα περίοδο προγραμματισμού αυξάνει και τα θετικά αποτελέσματα ελέγχου μας αποδεικνύουν ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Οι προσαρμογές που έγιναν ήταν οι σωστές και θα πρέπει να συνεχίσουμε έτσι, χωρίς να βιαζόμαστε να επιφέρουμε αλλαγές στο σύστημα. Ωστόσο, περαιτέρω απλοποίηση των προγραμμάτων και των διαχειριστικών συστημάτων επίσης επιβάλλονται, διότι η πολυπλοκότητα των ε, κανονισμών που ισχύουν σήμερα απαιτεί περαιτέρω δουλειά. Χρειάζεται ε, σε, ορισμένα μέτωπα οι κανόνες να γίνουν πιο απλοί, πιο κατανοητοί, ε, να εφαρμόζονται πιο εύκολα, αλλά και τα λειτουργικά προγράμματα, η χρηματοπιστωτική και μάλλον οικονομική διαχείριση για τις δημόσιες προμήθειες επίσης και αυτά χρειάζονται κάποια βελτίωση. Η πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού είναι θετικό μέτρο. Βέβαια, ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει τη μελέτη του θέματος αυτού το Συμβούλιο, ωστόσο, πολλά από τα θέματα που έχει επισημάνει το Ελεκτικό Συνέδριο το 2009 και πίσω, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στις διαπραγματεύσεις που θα έχουμε για τους νέους δημοσιονομικούς κανονισμούς. Αναμένουμε λοιπόν ε, τις συζητήσεις αυτές που θα γίνουν με τους εταίρους μας τους επόμενους μήνες. Επίσης, απλοποίηση πρέπει να γίνει στα επόμενα προγράμματα προκειμένου να οριστεί η νέα χρονική περίοδος. Σας θυμίζω όμως ότι η απλοποίηση ως κύριος στόχος δεν θα πρέπει να είναι σε βάρος της αποδοτικότητας των ελέγχων. Και τέλος, διαφανή αποτελεσματικά συστήματα για οικονομικές διορθώσεις. Και αυτό αφορά και την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις. Αυτοί οι μηχανισμοί είναι αναγκαίοι για να προστατεύονται τα συμφέροντα της Ένωσης σε σχέση με τους τελικούς δικαιούχους, οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αχρεωστήτως καταβλημένα κονδύλια θα πρέπει να επιστραφούν όταν υπάρχει απόδειξη ότι δαπανήθηκαν κακώς και η διακοπή των πληρωμών θα πρέπει να γίνεται αυθορή και παραχρήμα μόλις διαπιστωθεί μια παρατυπία επιπλέον ένα πλαίσιο όσον αφορά την αποτελεσματικότητα εκ μέρους Επιτροπής είναι ένα κίνητρο για να βελτιωθούν οι μηχανισμοί ανάκτησης στα κράτη-μέλη προκειμένου να αποφεύγεται οικονομική ζημιά. Έπειτα η διαφάνεια και ένας ε, αποτελεσματικός μηχανισμός διορθώσεων θα διασφαλίσει και τον πολίτη, τον Ευρωπαίο πολίτη και τον φορολογωμένο ότι τα χρήματα χρησιμοποιούνται σωστά με ύψιστη ευθύνη και αίσθημα υπολογίας. Και αυτό με φέρνει σε αυτό που είπα και στην αρχή, το θετικό μήνυμα προς τους Ευρωπαίους πολίτες, τώρα στον καιρό της κρίσης που ζούμε. Μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις για τον ετήσιο προπολογισμό το φετινό, το Συμβούλιο δεν θα πρέπει να ξαναδώσει την εντύπωση ότι ο προπολογισμό της Ένωσης έχει ξεφύγει από τη δυνατότητα διαχείρισης. Αυτό ήταν σε βάρος του κύρου όλων των θεσμικών οργάνων τη Ένωση, γιατί μόνο το Συμβούλιο είναι και το Κοινοβούλιο και για την Ένωση γενικότερα στο σύνολό τη. Πρέπει το μήνυμά μας να είναι σαφές, να στηρίζεται σε γεγονότα. Το ηλεκτρικό συνέδριο μας επιβέβαιωσε ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη δαπάνη της Ένωσης του 2009 βελτιώθηκε. Είμαστε στο σωστό δρόμο. Οι προσπάθειές μας πολιετής προσπάθειες αποδίδουν καρπούς και το μήνυμά μας για έναν καλύτερο μηχανισμό διαχείρισης των κονδυλίων έχει γίνει κατανοητό και από την Κομισιόν και από τις κυβερνήσεις. Το Συμβούλιο Εκοφήν της 15ης Φεβρουαρίου σημείωσε τις βελτιώσεις αυτές που αναφέρει το συνέδριο. Θυμίζοντα όλου του ενδιαφερόμενου, δηλαδή Επιτροπή Κυβερνήσει, ότι χρειάζεται περαιτέρω πρόοδο τα επόμενα χρόνια, τα αποτελέσματα του 2009 θεωρούνται ότι είναι θετικά, ότι υπόσχονται πολλά και σύσταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να δώσει την απαλλαγή στην Επιτροπή για την εκτέλεση του προπολογισμού 2009. Και πριν τελειώσω, θα ήθελα να αναφέρω τις συστάσεις απαλλαγής για τα διάφορα όργανα της Ένωσης που, έχουν, που είναι νομικά πρόσωπα και των οποίων η απαλλαγή προβλέπεται ω προ τον προπολογισμό της ένωση. Πολλά από του οργανισμού και οι αυτέ μπορούν ακόμα να βελτιώσουν την οικονομική του λειτουργία, όπω λέει και το Ελληνικό Συνέδριο, ωστόσο το Συμβούλιο κάνει σύσταση για απαλλαγή για όλε αυτέ τι υπηρεσίε. Επίση, απαλλαγή για τα έξι, έξι εκτελεστικά όργανα και υπηρεσίες και τι πέντε κοινέ υπηρεσίε με βάση τα DAS τα οποία έδωσε το Ελληνικό Συνέδριο. Κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σα. και είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν σχόλια, ερωτήσεις και διάλογο. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε ε, κύριε Υπουργέ. Όπως είπατε υπήρξατε πρώην συνάδελφος, τώρα μας μιλάτε ως υπουργό. Αυτό προϊονίζεται πολλά για περαιτέρω σύσφυξη των σχέσεων στην Ένωση. Κυρίες και κύριοι, θα επιτρέψουμε να δώσω το λόγο στον Επίτροπο κύριο Σεμέτα να μας πει την άποψη της Κομισιόν. Κύριε Επίτροπο, έχετε το λόγο. Ο Επίτροπος στα αγγλικά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, με κυρίε και κύριοι ευρωβουλευτές. Ήθελα να ευχαριστήσω την Ουγγρική Προεδρία του Συμβουλίου για τις ε, συστάσεις όπου ε, καλείται την αρμόδια αρχή για τον προπολογισμό να δώσει απαλλαγή για το 2009. Παρά τη σημαντική πρόοδο το 2009, παραμένουν ασθενή σημεία και χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά για όλους τους εμπλεκόμενους στη διαχείριση των προγραμμάτων της Ένωσης. Επιτροπή, κράτη-μέλη, που διαχειρίζεται περίπου το 80% του προπολογισμού. Πρέπει να βελτιωθεί η απόδοση στα δικά μας συστήματα ελέγχου. Τα καλύτερα συστήματα που έχουμε για τα νέα προγράμματα 2007-2013 θα λειτουργήσουν πλήρως μόνο αν εφαρμοστούν σωστά και από τις υπηρεσίες της Επιτροπής και από τις εθνικές αρχές. Δεύτερο, η οικονομική διόρθωση και η ανάκτηση των ποσών πρέπει να βελτιωθεί και η αναφορά προς την Επιτροπή θα πρέπει να γίνεται πιο έγκαιρα και με πιο αξιόπιστο τρόπο. Αυτό είναι σημαντικό προκειμένου να μειωθεί το ποσοστό σφάλματος και τα χρήματα της Ένωσης να φτάνουν σε αυτούς που τα χρειάζονται και για το σωστό σκοπό. Η Επιτροπή δεσμεύεται να συμβάλλει στις προσπάθειες αυτές προδραστικά όπου χρειάζεται, με προληπτικά εργαλεία και μέσα, διακοπή ενδεχομένως πληρωμών, παραδείγματο χάρη. Τρίτο, όλοι οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι πιο υπόλογοι όσον αφορά τα χρήματα του Ευρωπαίου Φορολογούμενου. Η διασφάλιση της Επιτροπής στο υπεύθυνο τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα κοινωτικά κονδύλια κράτη-μέλη και κάνουν αναφορά για αυτά. Η βελτίωση των δημοσιονομικών κανονισμών που λένε ότι οι εθνικέ αρχέ θα πρέπει να δώσουν μια ετήσια διαχειριστική έκθεση για όλα τα προγράμματα και με την κοινή διαχείριση. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το καλύτερο προκειμένου να έχουμε μια αξιόπιστη διασφάλιση ότι ο προπλογισμός της Ένωσης εκτελείται και ελέγχεται σωστά και ένα σημαντικό βήμα για βελτίωση της ε, στάσεις ευθύνης των κυβερνήσεων. Προσεχώς θα έχουμε συζητήσεις για την πρόταση αυτή. Θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα μάλιστα και σε ένα σεμινάριο που θα γίνει στις Βρυξέλλες με εκπροσώπους και από το Ευρωκοινοβούλιο, από το Συμβούλιο, από τις Εθνικές Αρχές και από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Και τέλος, η πολυπλοκότητα των κανόνων και των διαδικασιών είναι μια κύρια πηγή εσφάλματος. Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για μέτρα απλοποίησης σε σχέση πάντα με τους δικαιούχους. Τα μέτρα αυτά θα τα βρείτε στην αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού. Άλλα μέτρα θα τα βρούμε στη νομική βάση για τα προγράμματα επόμενων γενεών. Τελειώνω λέγοντας ότι η απαλλαγή για αυτό το έτος είναι μια ευκαιρία για όλους μας να επισημάνουμε τα, τα μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν αμέσως και μας δίνουν κατευθυντήρες γραμμές για την προσεχή δουλειά σε σχέση με την προετοιμασία των προγραμμάτων νέας γενιάς έτσι ώστε να υπάρξει η σωστή προστιθέμενη αξία και τα χρήματα να χρησιμοποιούνται με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε μέτα Τρεις ομιλητές έχουν ζητήσει το λόγο. Πρώτα οι συντονιστές των πολιτικών ομάδων και μετά οι βουλευτές. Κανείς συντονιστής δεν θέλει το λόγο. Ο κύριος Χατζημαρκάκης παρακαλώ. Ως συντονιστής. Και ως εισηγητής ε, ελαφρώς θα ήθελα να λάβω το λόγο. Ε, μα στο σημείο 7 είναι το θέμα σας. Εσείς θέλετε να μιλήσετε από τώρα. Ναι, θέλω να μιλήσω και από τώρα. Καλώς. Παρακαλώ. Περιμένετε τη σειρά σας όμως, γιατί πρώτα είπαμε οι συντονιστές. Ο κύριος Φιέλνερ. Κύριε Χατζημαρκάκη, τέταρτο στη σειρά είστε. Ο κύριος Φιέλνερ. Τώρα έχω μπερδευτεί. Έχουμε διάφορα θέματα, διάφορα σημεία στην μέση διάταξη που είναι αλληλοεπικαλυπτόμενα. Να κάνω λοιπόν ερώτηση τότε. Στον αξιότιμο κύριο Υφυπουργό και να επικεντρωθώ εγώ στο Συμβούλιο τότε αυτά που συστήνει το Συμβούλιο για την απαλλαγή. Και στη συνέχεια θα επανέλθω στην έκθεση του κυρίου Χατζημαρκάκη και ε, στον Επίτροπο. Καλό σας φαίνεται αυτό. Ωραία. Γιατί έχω μπερδευτεί λίγο. Λοιπόν, ε, ήταν ε, ενδιαφέρον να σας ακούει κανείς και να ακούει και τι διαδίδεται για τη συζήτηση στο Συμβούλιο. Θα ήθελα να ακούσω κάποιο σχόλιο του Συμβουλίου, γιατί από ό,τι έμαθα, δεν ήταν ομόφωνη η απόφαση. Τρία ήταν τα κράτη-μέλη τα οποία αυτή τη φορά απήχαν. Και εξ όσων γνωρίζω αυτό είναι πρωτοφανέ. Πώς γίνεται αυτό, για ποιο λόγο έγινε, μπορείτε να μας το σχολιάσετε λίγο. Κάντε μας μια δήλωση, όχι ως Προεδρία βέβαια, αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να τα ακούσουμε. Κάτι άλλο επίσης ενδιαφέρον, σχόλιο από πλευρά σας, για τις δηλώσεις αξιοπιστίας των κρατών μελών, για τον τρόπο με τον οποίο εκτελούν τον προπολογισμό. Αυτό το συζητήσατε στο Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της συζήτησης απαλλαγή. Γιατί γνωρίζουμε ότι και σωστά επισημάνατε υπάρχουν τομεί, όπως είναι τα διαρθρωτικά ταμεία, το περιφερειακό ταμείο που υπάρχουν αδυναμίες. Και εδώ στο Κοινοβούλιο, εδώ και καιρό συζητούμε ε, για την υπόθεση αυτή και ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να το κάνουν κτήμα του και να αισθάνονται ευθύνη για αυτό το θέμα. Το έχετε συζητήσει αυτό, τις εθνικές ε, ε, δηλώσεις διαχείρισης και πώς μπορείτε να βοηθήσετε εκεί για ένα καλύτερο έλεγχο τη διαχείριση των κονδυλίων. Αυτέ τι ερωτήσει θα ήθελα να κάνω εγώ στον Υφυπουργό τη Ουγγαρία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να απαντήσει πρώτα ο Υφυπουργό, μάλλον όχι. Πρώτα να ομαδοποιήσουμε τι ερωτήσει σα και στη συνέχεια θα απαντήσει ο Υπουργό. Ο κύριος Ζόντεργκαρτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό για τι ε, ερωτήσεις του. Εγώ έχω να κάνω τρεις, για τι απαντήσει, συγγνώμη. Έχω να κάνω τρεις ερωτήσεις. Υπογραμμίσατε κάποιες βελτιώσεις που έγιναν σε ορισμένου τομεί. και αν κατάλαβα καλά, δηλώνεται ότι είναι βελτίωση η μείωση του σφάλματος από 11% σε 3%. Για μένα η βάση είναι οι νέοι κανόνες. Ε, δηλαδή αυτό τι σημαίνει, ότι με τους νέους κανόνες τώρα αποκλείεται το στατιστικό σφάλμα, ε, το τυχαίο σφάλμα δηλαδή, για λόγους στατιστικούς. Του χρόνου περιμένετε επιδείνωση, η πραγματική υποχώρηση. Γιατί εάν βελτιώθηκε η κατάσταση λόγω των κανόνων, ε, θεωρώ και, και τον επόμενο χρόνο θα βρίσκουν εφαρμογή οι κανόνες αυτοί, καθότι είναι μόνιμοι και διαρκείς. Λοιπόν, για το επόμενο έτος ε, έχετε αισιόδοξη στάση, είναι μόνιμη συμβελτιώσει συνεχή. Στη συνέχεια, τι είπε το Συμβούλιο για τη μεγαλύτερη ευθύνη των κρατών. Έχει θέση από αυτού. Ακούμε δηλώσεις των Υπουργών ε, Οικονομικών για την αύξηση ακριβώς των ευθυνών των κρατών. Ένα τρίτο που συζητούμε και είναι καλό είναι οι περιφερειακοί οργανισμοί, agencies, ε, θέματα τη διαχείριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εδώ στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού θέλουμε συγκεκριμένε απαντήσει στι ερωτήσει που θέτουμε. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω αν μπορεί ο κύριο Υπουργό να μα απαντήσει σε αυτό και στι ερωτήσει που θέτουμε εμεί στο Συμβούλιο. Σα ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ιβάνοφ. Ε, θα, ε, ναι, ναι, θα έχουμε συνδυασμένες ερωτήσεις και μετά... Ε, εγώ έχω ερώτηση για την γενική συζήτηση, όχι για τον Υπουργό. Έχουμε άλλες ερωτήσεις. Τότε θα δοθούν οι απαντήσεις. Ο κύριος Χατζημαρκάκης όμως. Α, συζήτηση ή ερώτηση. Ε, μπορώ να θέσω 100 ερωτήσεις, αλλά θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Προεδρία του Συμβουλίου για το ανοιχτό πνεύμα, διότι είσαστε πάρα πολύ ανοιχτός και βλέπουμε επίσης, διαπιστώνουμε μια αλλαγή. Αλλά, ωστόσο, θα πρέπει να πω στο Συμβούλιο ότι υπάρχει κάποια σχιζο... είναι κάπως σχιζοφρενικό αυτό που μας παρουσιάζεται, διότι από τη μία πλευρά έρχεται εδώ ε, με το καπέλο του Συμβουλίου ενός Ευρωπαϊκού Θεσμικού Οργάνου που ως ορισμένο σημείο επιτίθεται σε, ως ένα ορισμένο σημείο, σε ένα ορισμένο βαθμό, επιτίθεται στην Επιτροπή και βλέπετε ότι είσαστε πιο νόμιμοι, πιο, έχετε περισσότερη νομιμότητα, κανονικότητα, το διαβάζουμε αυτό και από την άλλη πλευρά εσείς, εσείς και τα κράτη-μέλη έχετε το πρόβλημα να συμμορφωθείτε προς τους κανόνες που ζητάτε να τηρήσει η Κομισιόν. Το, πιο, το παράδειγμα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι μεταξύ των τριών χωρών που δεν ε, συνυπέγραψαν ε, το ψήφισμά σας, απήχαν και αυτό είναι καινούριο και για πρώτη φορά κράτη-μέλη απήχαν οι κάτω η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, διότι δεν είναι υπέρ της κατάστασης ε, της κατάστασης διαχείρισης των κονδυλίων και από την άλλη πλευρά στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, είχαμε όλα τα προγράμματα που διακόψαν το 2010. Και θέλω να σας ρωτήσω τι επιδιώκετε, τι, σε τι αποβλέπετε. Μπορώ να σας πω ότι μετά από 16 χρόνια όπου εσείς είπατε ότι δεν υπάρχει θετική ντάς ε, δήλωση συμμόρφωσης και αξιοπιστίας, ζητάτε λεπτομέρειες για να δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα και πρέπει να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Σεμέτα που, ήταν, που επέδειξε πνεύμα συνεργασίας για να κάνουμε ένα πράγμα, διότι έχουμε μόνο ένα όπλο για να είμαστε ειλικρινείς ε, κατονομάζοντας τα κράτη-μέλη που συνεργάζονται και κατηγορώντας τα κράτη-μέλη που δεν συνεργάζονται. Έχουμε λοιπόν το Ηνωμένο Βασίλειο που από τη μια πλευρά μας επιτίθεται, ζητάει περισσότερη διαφάνεια, συμμόρφωση προς την κανόνα και η ίδια, η χώρα δεν συμμορφώνεται προς τους κανόνες. Τι σχιζοφρενική τακτική είναι αυτή ε, διότι έχουμε μια κρίση εμπιστοσύνης και οι φορολογούμενοι θέλουν εμείς και εσείς ως πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και χαίρομαι που είστε εδώ μεταξύ μας διότι καταλαβαίνετε την δική μας θέση. Εμείς μπορούμε να απευθυνθούμε μόνο στην Επιτροπή. Αλλά η Επιτροπή έχει δυσκολίες να αποδώσει αποτελέσματα διότι όπως είπατε 80% των κονδυλίων έχουν κοινή διαχείριση. Τα κράτη-μέλη λοιπόν δεν επιδεικνύουν σαφή διαφάνεια και επανέρχομαι στην ερώτηση του κυρίου Πιάνος για την δήλωση εθνικής διαχείρισης. Τα περισσότερα κράτη-μέλη ε, δεν παραδίδουν ουσιώδεις πληροφορίες για το πώς γίνεται η διαχείριση των δαπανών. Αυτό που έχουμε επιτάπτωσα ε, και ο κ. Σεμίτας δεν αναφέρθηκε άμεσα αλλά στην συνεργασία που έχουμε

Ε, με την Κοκομπιού εργαζόματα πάνω σε αυτό. Η Κομισιόν θα σας ζητήσει τουλάχιστον μια δήλωση σε διοικητικό, διαχειριστικό επίπεδο. Ε, δεν θα υπογράψουν οι Υπουργοί όπως ε, ζητάει τώρα εδώ και πέντε χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά θα είναι μια δήλωση σε διοικητικό επίπεδο. Έχουμε πέντε κράτη που έχουν δώσει πολύ ουσιαστικές πληροφορίες, ένα κράτος ή κάτω χώρες πολύ καλές πληροφορίες και όλοι οι άλλοι είμαστε 27 μέλη που δεν δεν μας δίνουν τίποτα. Δεν παραδίδουν τίποτα, δεν υποβάλλουν. Πώς λοιπόν από τη μία πλευρά οι δηλώσει σας είναι τελείως αποδεκτές, ε, συμμορφώνονται με τα όσα λέμε εμείς ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά εμείς δεν διαχειριζόμαστε τα κονδύλια, εσείς τα διαχειρίζετε και στα 30% για το Ταμείο Συνοχή, 40% το ελεγκτικό συνέδριο μας λέει και το πιστεύουμε αυτό ότι όλα τα προβλήματα, όλα τα σφάλματα μπορούσαν να ανοιχνευτούν πριν από τις δαπάνες, από την εκτέλεση των δαπανών. Ποια είναι η πραγματική σας στρατηγική, διότι εσείς δηλώνετε ότι εδώ δεν έχουμε ε, θετική τάση, έχουμε αρνητική δήλωση αξιοπιστίας, έχουμε απαλλαγή. Πώς θα γίνει αυτό και τι μπορεί να βελτιωθεί για να τεθεί τέρμα στην σχιζοφρένεια, διότι πρόκειται για σχιζοφρενική κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο αν θα κάνει ερώτηση ή θα κάνει μια γενική παρατήρηση. Αν είναι ερώτηση θα την απαντήσουμε, αλλά αν δεν είναι ερώτηση... Είναι περίπου τέτοιες ερωτήσεις ε, σαν αυτές που έθεσε και ο εισηγητής ο ίδιος, διότι... Καταρχάς, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον κύριο Υφυπουργό για τις δηλώσεις του Συμβουλίου. Η πρώτη πρόταση που σημείωσα είναι ότι το Συμβούλιο ανησυχεί. Μπράβο, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Και εμείς ανησυχούμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Διότι η συμπεριφορά του Συμβουλίου και των κρατών μελών όταν πρόκειται για θέματα οικονομικά, για μένα τουλάχιστον, είναι όλο και λιγότερο κατανοητή. Δεν καταλαβαίνω τη συνέπεια ούτε τη στάση του Συμβουλίου σε θέματα δημοσιονομικά και οικονομικά. Τα τελευταία χρόνια, όταν συζητούσαμε για το προπολογισμό του 2011, συγκεκριμένα πέρυσι, συζητούσαμε νύχτε ολόκληρε με εκπροσώπου των κρατών μελών για μελλοντικές χρηματοδοτήσεις και διαχείριση και νύχτε επίση ολόκληρε για το πώ θα πρέπει να διαμορφωθεί ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα κάνω με την ιδιότητα ως ε, υπεύθυνο για τον προϋπολογισμό. Ως υπεύθυνο όμως για τον έλεγχο του προϋπολογισμού έχω την ίδια εμπειρία με τον κύριο Χατζημαρκάκη. Μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει βλέπουμε κράτη-μέλη να ε, μη διαχειρίζονται παρκώς ε, τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διοικητικό επίπεδο και είναι τα ίδια κράτη-μέλη που λένε κανονικά θα πρέπει να μειωθεί ο προπολογισμό. Σας ερωτώ, έπαιξε αυτό κανένα ρόλο κύριε Υπουργέ στο ΕΚΟΦΗΝ. Το Συμβούλιο συζητάει αυτά τα θέματα με τα κράτη-μέλη. Διότι πιστεύω ότι και στην απαλλαγή, εάν κάποια κράτη θέλουν να ψηφίσουν αποχή, αυτό σημαίνει ότι κάνουν ουσιαστικά πρόταση μορφής στον ίδιο του στον εαυτό, γιατί τα κράτη διαχειρίζουν τα χρήματα. Και τι γίνεται με τα συστήματα διαχείρισης. Υπάρχουν τα εξή δύο φαινόμενα. Ε, ομολογώ ότι είναι πάρα πολύ περίπλοκο το σύστημα ε, στις γεωργικές δαπάνες, που όμως έχουμε φτάσει σε επίπεδα σφάλματος αποδεκτά με το σύστημα αυτό. Ταυτόχρονα όμως το ελεγκτικό συνέδριο στην ετήσια έκθεση μας κοινοποιεί ότι ένα τμήμα των συστημάτων που είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, γιατί το λέει και η συνθήκη αυτορυτά, ε, λειτουργεί με τρόπο ανεπαρκή. Λοιπόν, τα ίδια κράτη-μέλη έρχονται και λένε θα πρέπει να γίνεται πιο χρηστή διαχείριση και πιο καθαρή. Ναι, ωραία. Εδώ παραβιάζεται ανοιχτέ θύρε στο Κοινοβούλιο, συμφωνούμε και επαυξάνουν. Αλλά τα κράτη-μέλη τι κάνουν για να ανταποκριθούν στι ίδιε του τι απαιτήσει και να τι εφαρμόσουν. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Η Νέσα Γιάλα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν μπορώ να μην μπω στον πειρασμό ε, να μιλήσω <laughs> κι εγώ γι' αυτό. Καλωσορίζω τον κύριο Μπέξη από την άλλη πλευρά του λόφου και το συγχαίρω για το διορισμό του. Θα ήθελα κι εγώ, αν γίνεται, να μας μιλήσετε λίγο για αυτό το θέμα. Το Συμβούλιο δηλαδή πώς βλέπει τα πράγματα και πώς το βλέπει η Ουγγρική Προεδρία που μπορεί να έχει όλες τις καλές προθέσεις αλλά μέχρι τώρα το Συμβούλιο το ίδιο δεν καταφέραμε να ανταποκριθεί στα αιτήματά μας σε ό,τι αφορά την έγκριση και την απαλλαγή για τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Δεν είμαστε στο επίπεδο που ήμασταν πέρσι επί Ισπανικής Προεδρίας. Είχαμε φτάσει σε μια συμφωνία πλέον τέτοια εποχή πέρυσι. Καθόλου δεν αφισβητώ τις καλές προθέσεις, επαναλαμβάνω και την προθυμία της Ουγγρικής κυβέρνησης. Αλλά τι γίνεται με το Συμβούλιο και τη διαχείριση των θεμάτων εκεί. Ε, θα σας παρακαλούσα να μας πείτε τι γίνεται με τα έγγραφα. Γιατί ούτε καν ε, στην απάντηση των ερωτημάτων μας στη γραπτή δεν ανταποκρίθηκαν, πράγμα που πέρσι είχε λυθεί τέτοιο καιρό. Εμείς πώς να κινηθούμε αν δεν βλέπουμε συγκεκριμένα απτά χειροπιαστά αποτελέσματα πριν από οποιαδήποτε συνάντηση, συνεδρίαση, για να μην πω συνδιαλλαγή. Ευχαριστώ. Thank you very much. And now I'd like to ask Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκρέσλε. θέλω να πω για τη συζήτηση μετά, λέγε. Κυρία Γκρέσλε. Δεν ήθελα το λόγο για αυτό το θέμα τώρα, για τη γενική συζήτηση μόνο. Γιατί θεώρησα ότι οι σκιώδεις ηγητές μας θα μιλήσουν προηγουμένως. Ναι, μιλήσαμε, λέει ο κύριος Φέλνερ. Α, μάλιστα. Καλά. Έχω άλλη ερώτηση. Γιατί έχουμε και άλλο εργοτάξιο με το Συμβούλιο και αυτό είναι η απαλλαγή του Συμβουλίου, του ίδιου. Και θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται εκεί και πώς θα προχωρήσουμε και ποιες είναι οι θέσεις. Γιατί λέει προετοιμάζουν ένα memorandum of understanding που θα μπει λέει την Τετάρτη ε, στο Κορεπέρ Πιο understanding. Ε, βλέπετε καμία συνεννόηση πουθενά για να κάνουμε και μνημόνια συνεννόησης μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Ε, τα δημοκρατικά μας δικαιώματα θα περισταλούν κατά πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν κατάλαβα. Ε, ε, με το ίδιο πνεύμα προχωράει το Συμβούλιο και σε αυτή την απαλλαγή. Στη Γερμανία γίνεται μεγάλη συζήτηση αυτό τον καιρό για το διδακτορικό ενός υπουργού που τον ονομάζουν τώρα Υπουργό Copy-Paste, αντιγραφέας. Ε, και αν δούμε και το θέμα της απαλλαγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πάλι τα ίδια ισχύουν. Και το θέμα δεν είναι να αλλάξουμε μόνο το χρόνο, τη χρονιά και το οικονομικό έτος και κάπως να προσαρμόσουμε τα στοιχεία. Νομίζω ότι το Συμβούλιο είναι πολύ μεγαλόθυμο με τον εαυτό του και υπάρχει και μια σύγκρουση συμφερόντων. Και η σύγκρουση συμφερόντων είναι κάτι το οποίο απασχολεί το Συμβούλιο και πώς το αντιμετωπίζετε στο Διενικές. Πότε σκοπεύετε να έχετε μια πρόταση για να ελπίζουμε ότι θα βελτιωθεί η εκτέλεση των προγραμμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχω ακόμα έναν ομιλητή. Ομιλήτρια την κυρία Ιβάνοβα. Δεν ξέρω αν θέλει το ελεγκτικό συνέδριο να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Ιβάνοβα, έχετε το λόγο. Θα ήθελα να σχολιάσω περισσότερο σε σχέση με την Επιτροπή, απαλλαγή της Επιτροπής. Εφόσον έχουμε εδώ την ευκαιρία να θέσουμε ερωτήματα στην Προεδρία, Παρόλο που τα περισσότερα σε ερωτήσει έχουν τεθεί, θα ήθελα παρόλα αυτά να ρωτήσω τι μπορείτε να κάνετε εσείς ως ε, Προεδρία για το ε, θέμα των ε, δηλώσεων εθνικής διαχείρισης και επιφυλάσσομαι να παρέμβω αργότερα με σχόλια για την Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Γαρμπράντη. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω μια, μια πολύ σύντομη ερώτηση. Ένα από τα ουσιώδη στοιχεία της δημοκρατίας είναι η πολιτική υπευθυνότητα και η πολιτική λογοδοσία. Ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα 16 έτη που δεν έχουμε πραγματική πολιτική λογοδοσία η ερώτησή μου στον ε, Υφυπουργό που εκπροσωπεί τα 27 κράτη-μέλη εδώ είναι η εξής. Πώς είναι δυνατόν ένα, μια τέτοια ε, θεμελιώδης αξία της δημοκρατίας, η πολιτική υπευθυνότητα και λογοδοσία ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να μην υπάρχει, να μην υπάρχει από τα κράτη-μέλη, γιατί ακόμα απομακρύνονται, παρεκκλίνουν, αποφεύγουν την πολιτική τους υπευθυνότητα. Βρίσκω τόσο δύσκολο να εξηγήσω σε κάποιον πάνω σε αυτόν τον πλανήτη ότι τα κράτη-μέλη δεν αναλαμβάνουν την πολιτική τους ευθύνη. Ε, δεν μιλάω για διαχειριστικές δηλώσεις, διότι για να μην ειλικρινής δεν, μας, δεν με ενδιαφέρουν. Έχουμε ένα πολιτικό σώμα, ελέγχουμε άλλες ε, πολιτικές οντότητες. Μπορείτε να απαντήσετε στην ερώτηση αυτή για μένα. Ευχαριστώ κύριε Κομπρά εξ ονόματος του ελεγκτικού ε, συνεδρίου, κυρία Καριουλάιτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως, το ελεγκτικό συνέδριο δεν θέλει να αρχίσει μια πολιτική συζήτηση, αλλά δράτω με τις ευκαιρίες λέγοντας ότι το συνέδριο ε, είναι ε, ε, ικανοποιημένο που μπόρεσε να συμμετάσχει στην συζήτηση για τον προϋπολογισμό 2009 και να έχει έκθεση και οι συστάσεις έχουν υιοθετηθεί. Δεν έχουμε ε, καμία, κανένα πρόβλημα με την ερμηνεία των εσωτερικών λογιστικών ελέγχων, αλλά θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις τα επόμενα χρόνια για να δούμε αν η τάση αυτή θα διατηρηθεί. Ε, και είχαμε και ορισμένε παρατηρήσει σχετικά με την προσέγγιση ως προς τον λογιστικό έλεγχο. Σα ευχαριστώ για αυτήν την συνεκτική παρέμβαση. Κύριε η κυρία Μακοβέη. θέλετε πάρα πολύ να λάβετε τον λόγο ή δεν θέλετε, διότι δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Η δεν θελετε διοτι δεν εχουμε παρα πολυ χρονο τη γραμματεια μου, λέει, μου είπε ότι θέλατε να λάβετε τον λόγο. Θέλετε ακόμη να λάβετε τον λόγο. Διότι πιέζει ο χρόνος. Θα ήθελα να θέσω ερωτήσεις όταν ε, συζητήσουμε την απαλλαγή σχετικά με την Επιτροπή. Νομίζω ότι είναι το επόμενο σημείο. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, εάν μπορώ να σας ζητήσω να προσπαθήσετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις αυτές. Έχουμε 10 λεπτά για αυτό. Αν μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας ε, την εμπειρία σας. Ε, τι σημαίνει να αλλάζει κανείς παπούτσια, να έρθει εδώ εκ μέρους ε, της, του Συμβουλίου σε σχέση με τον προηγούμενο ρόλο σας ως μέλος αυτού του Κοινοβουλίου. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να αναφερθώ στην ερώτησή σας. Πραγματικά ο ρόλος άλλαξε. Γιατί θυμάμαι νομίζω ήμασταν μαζί στην Επιτροπή Μεταφορών που είχαμε μια πάρα πολύ γόνιμη συνεργασία από κάθε άποψη. Όταν όμως ε, μπει σε έναν άλλο ρόλο και μην ξεχνάμε ότι είμαστε 27 χώρες μέλη και μερικά είναι ίσα, ισότιμα μεταξύ του, μερικά πιο ισότιμα από τα άλλα. Είναι ένα σημαντικό ερώτημα δηλαδή αυτό στο οποίο αναφερθήκατε. Πάντω είναι ε, πολύ ευγενέ εκ μέρου σα ότι αναφερθήκατε σε αυτό και ελπίζω να είμαι στο ύψο των περιστάσεων. Πολύ σύντομα λοιπόν απαντώ ω εξή. Αποχή στο Συμβούλιο. Όντω, τρει χώρε δήλωσαν αποχή στο Συμβούλιο και ίσως όλοι ξέρετε ότι δέχτηκαν όχι να μονόπλευρες δηλώσεις, αλλά εφιστώ την προσοχή σας στο ότι το 85% των ψήφων στο Συμβούλιο ήταν υπέρ και 24 κράτη-μέλη. Άρα ουσιαστικά η πλειοψηφία στο Συμβούλιο συμφώνησε με τα πορίσματα του Συμβουλίου και στην Κορεπέρ και στην ε, Επιτροπή Προπολογισμών του Συμβουλίου. Οι τρεις χώρες που έκαναν αποχή δεν καταψήφισαν το επισημένο αυτό. Ο πρόεδρος ζητάει, ζητάει ονόματα. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω την έγκριση που χρειάζεται να πω ποιες είναι οι χώρες αυτές. Είπα τρεις χώρες. Η ερώτηση είναι σαφής και υπολογίζουμε και τα κράτη-μέλη που ε, επισημαίνουν ότι έχουν εσωτερικές διαδικασίες οι οποίες είναι πιο δεσμευτικές σε σχέση με τους διαχειριστικούς κανόνες και εν γέννη τους κανόνες της Ένωσης. Ωστόσο, ακόμα και αυτές οι χώρες μέλη ε, δέχτηκαν τα ελεγκτικά πορίσματα του συνεδρίου και είπανε ότι θέλουν να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στη διαχείριση των κονδυλίων και για το 2009. Αυτό αναφέρεται στο κείμενο. Αλλά στις προσεχείς διαπραγματεύσεις, και αυτό είναι το πολιτικό νομίζω μήνυμα το, πιο σημαντικό για την διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση του, του κανονισμού, θα είναι μια ευκαιρία για όλους. Επιτροπή, Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κυβερνήσεις να τα ξαναδούνε όλα αυτά τα θέματα τα οποία ετέθησαν. Πάντως η διαχείριση βρίσκεται όπως είπα στο σωστό δρόμο. Όσον αφορά την πολιτική ευθύνη, κάποιος συνάδελφος ανάφερε το σημείο αυτό. Και έχει δίκιο. Όλοι έχουμε πολιτική ευθύνη. Αλλά η συνθήκη ορίζει ότι την πολιτική ευθύνη την έχουν τα θεσμικά όργανα. Το Συμβούλιο, το Ευρωκοινοβούλιο. Το Συμβούλιο, η πολιτική του ευθύνη σχετίζεται με την τήρηση της συνθήκης της Λισαβόνας. Εμείς ασκούμε την πολιτική μας αυτή ευθύνη και ως προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ως προς το Συμβούλιο φυσικά με το να ακολουθούμε και να τηρούμε τους κανόνες. Δηλαδή να παίρνουμε την έκθεση του Συναδρίου, να την αναλύουμε και να δούμε αν με βάση τα απορίσματα αυτά του συνεδρίου τι σημειώθηκε. Βελτίωση και τι επιπλέον βελτιώσεις μπορούμε να κάνουμε με αντίστοιχα μέτρα. Είχαμε σημαντική βελτίωση σχετικά με τη μείωση του ποσοστού σφάλματος. Και γι' αυτό είπα ότι είμαστε σε σωστό δρόμο και σωστό είναι να ξεκολουθήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Βέβαια και οι κυβερνήσεις και ο έλεγχος στα κράτη-μέλη και αυτόν ο ρόλος είναι σημαντικός. Αλλά αυτό είναι θέμα των κυβερνήσεων να στραφούν προς τους ψηφοφόρους και να δουν. Υπήρξε παρατυπία, έγινε ανάκτηση, υπήρξαν αρνητικές κυρώσεις ή αρνητικές συνέπειες γενικότερα. Να στραφούν λοιπόν προς τους εκλογείς τους και να κάνουν αυτούς τους συλλογισμούς. Άλλο σημαντικό θέμα είναι ο μηχανισμός απαλλαγής του Συμβουλίου. Αν και εγώ έχω έρθει εδώ να σας μιλήσω για τον μηχανισμό απαλλαγής της Κομισιόν, αυτό είναι το θέμα στην ημερήσια διάταξη σήμερα, με βάση τη συνθήκη, και το ξαναλέω αυτό, εγώ εκπροσωπώ και την κοινή θέση του Συμβουλίου, αλλά και το πνεύμα και το γράμμα της συνθήκης και δίνουμε την απαλλαγή για το σύνολο του προπολογισμού του 2009 για την Επιτροπή. στη διαχείριση του προπολογισμού. Παρ' όλα αυτά, θα θέλαμε πρόοδο και για άλλες μορφές συνεργασίας αν και με βάση την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου και με βάση εσωτερικέ εκθέσεις δεν υπάρχουν ειδικέ παρατυπίες σχετικά με την διαχείριση της διοίκησης και αυτό ισχύει για όλα τα θεσμικά όργανα, Συμβούλιο, Ευρωκοινοβούλιο, Επιτροπή. Προκειμένου όμως να έχουμε μια καλή συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωκοινοβουλίου θα θέλαμε να σημειωθούν περαιτέρω βήματα. Και πιστεύω στις επόμενες εβδομάδες ως συνέχεια της θέσης του Κοινοβουλίου σύντομα ελπίζω να έχουμε μια προσφορά προς το Ευρωκοινοβούλιο για συμφωνία. Γιατί η συμφωνία μπορούμε να το πούμε ένα μνημόνιο κατανόησης. Η κυρία Γκρέσλε είπε ότι δεν υπάρχει κατανόηση ή συμφωνία μεταξύ μας. Πρέπει όμως να υπάρχει συμφωνία, διότι αν κάτι δεν το ρυθμίζει η συνθήκη και θέλουμε να σημειωθεί η πρόοδος, βάσει την καλή προαίρεση μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων χρειαζόμαστε ένα μνημόνιο, στο πούμε, κοινή συνεννόηση περί του πρακτέου. Αν αναλάβουμε τις ευθύνες μας, εμείς, εσείς, και επειδή υπήρξα ευρωβουλευτής επί πέντε χρόνια, γνωρίζω πόσο απόλυτα νόμιμος είναι ο ρόλος του Ευρωβουλευτή στο σημείο αυτό. Πρέπει να υπάρξει αυτή η συμφωνία, επαναλαμβάνω, με βάση τα ίσα δικαιώματα και την ισοτιμία μεταξύ των θεσμικών, θεσμικών οργάνων μας και πιστεύω ότι μπορεί να επιτευχθεί αυτό τις επόμενες τις προσεχείς εβδομάδες. Αυτά είχα να σας πω και πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε με αυτό το πνεύμα. Και όταν μιλάμε για πολιτική ευθύνη θα θέλω να αναφέρω και κάτι άλλο που είναι σημαντικό. Μη συνδέουμε θέματα όπως η απαλλαγή του 2009 με άλλα θέματα. Και σας παρακαλώ να μην συνδέετε θέματα γιατί το πιο σημαντικό τους επόμενους μήνες είναι να σημειωθεί ένα θετικό βήμα σε σχέση με την απαλλαγή του 2009 και παράλληλα η συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων που εκπροσωπούμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Χρειάζεται ευελιξία από όλε τι πλευρέ, από τι δύο πλευρέ εν προκειμένου, προκειμένου να πετύχουμε ένα σωστό αποτέλεσμα. Ξέρω ότι δεν έχω χρόνο κύριε Πρόεδρε όπω μου το επισημαίνετε. Ο Πρόεδρος λέει έχετε ακόμα τέσσερα ολόκληρα λεπτά. Ήταν πιο εύκολο όταν ήμουν ευρωβουλευτή, λέει ο υπουργό. Ίσως αργά ή γρήγορα ξανατεθεί το θέμα αυτό. Λοιπόν, για το Ταμείο Συνοχής και την διαχείρισή του όπως σας είπα, το 2009 ήταν η πρώτη χρονιά που το Ελεκτικό Συνέδριο ε, ανάλυσε τις ε, ε πληρωμές 2009 και μετά για το Ταμείο Συνοχής. Ελπίζω να συνεχιστεί αυτό. Και ζητήσαμε και από τα κράτη-μέλη να έχουν διατάξεις ελέγχου πιο αυστηρές σε σχέση με τα αποτελέσματα των δικών μας ελέγχων. Οι αιτήσεις ε, συνόψεις και οι συνθετικές εκθέσεις είναι χρήσιμες προκειμένου να έχουμε διαφάνεια στην εκτέλεση του προπολογισμού. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Όμως, δεδομένη της πρότασης της Επιτροπής για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού, ελπίζω να υπάρξει ένα ακόμα πιο σημαντικό βήμα στη διαδικασία αυτή. Μια πιο διαφανή και απλουστευμένη διαδικασία για τον έλεγχο. Και βέβαια είναι και η κρίση οικονομική, αλλά το θέμα είναι μέχρι σε ποιο βαθμό θα πρέπει να φτάσουμε, ποιο είναι ο βέλτιστος βαθμός για να έχουμε και μεγαλύτερο έλεγχο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Θα πρέπει και αυτό να το λάβετε υπόψη. Ωστόσο, Αυτό που θέλω να πω είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για τέτοια θέματα είναι ότι έχει προστιθέμενη αξία. Έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν τέτοια ζητήματα, τα έχουμε εξετάξει, αλλά θα επανέλθω τις επόμενες εβδομάδες στο θέμα αυτό. Τώρα, για την απαλλαγή του Συμβουλίου νομίζω αναφέρθηκα ήδη σε αυτή. Αν δεν απατώμε, τι άλλο με ρωτήσατε. Μάλιστα. Καταλήγω, γιατί έχω ένα λεπτό μόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για ε, τις απόψεις σας, τα έχω σημειώσει. Σημειώνω ότι Συμμεζόμαστε πολλέ ανησυχίε και θα τα πω αυτά στο Κορεπέρ, στην ε, Επιτροπή που χειρίζεται τα θέματα του προπολογισμού και είναι σημαντικό ε, να συνεργαζόμαστε όλοι μαζί επικοδομητικά όλα τα θεσμικά όργανα για μια χρηστή οικονομική διαχείριση και σωστή εκτέλεση του προπολογισμού και να στείλουμε καλό μήνυμα στον Ευρωπαίο φορολογούμενο πολίτη. Το λέει και το ελεγκτικό συνέδριο ότι βελτιώθηκε η διαχείριση των κοινωτικών πόρων και το ξαναλέω, βελτιώθηκε. Μα ενθαρρύνει αυτό να προχωρήσουμε προ τα εμπρό στον ίδιο δρόμο που στην κατεύθυνση αυτή. Αγαπητά μέλη, αγαπητοί συνάδελφοι ή πρώην συνάδελφοι για να σα λέω έτσι, ελπίζω τι επόμενε εβδομάδε να ε, έχουμε καλές συζητήσεις και για τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για το Δημοσιονομικό Κανονισμό και για την εμβάθυνση των θεμάτων αυτών, αλλά και στο παρόν πλαίσιο θα ήθελα να σας ζητήσω να αναλάβετε και εσείς την ίδια σας την πολιτική ευθύνη και θετική ε, στάση να δείξετε ε, στην απαλλαγή του 2009. Αυτά ήθελα να σας πω γιατί ο χρόνος μου τελείωσε και ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Πολύ εντυπωσιακά αυτά που μας είπατε. Η κυρία Ινέσα Γιάλα Α, θέλει να σας κρατήσει άλλα 40 δεύτερα, δεν σας αφήνει να φύγετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, πάρα πολύ σύντομα. Ευχαριστώ τον κύριο Μπέξη για τις εξηγήσεις του, για την απαλλαγή του Συμβουλίου. Το ξέρω ότι δεν είχε προβλεφτεί η συζήτηση, αλλά δεν μπορούσα να αντισταθώ στον πειρασμό, να μην το αναφέρω. Και θέλω να σας πω ότι ακριβώς επειδή έχουμε ευθύνη εμείς και είμαστε υπεύθυνοι για την απαλλαγή, εμείς είμαστε ε, οι, ε, αρχή που φέρει την ευθύνη να το εγκρίνουμε το θέμα της απαλλαγής, όχι συστάσεις. Δεν κάνουμε συστάσεις. Εμείς εγκρίνουμε. Εμείς είμαστε η αρμόδια εκείνη αρχή για την έγκριση ή και τη μία έγκριση της διαχείρισης. Δεν κάνουμε εμείς συστάσεις. Ξέρουμε ότι οι συστάσεις είναι άλλου είδους ευθύνη. Εμείς φέρουμε την τελική ευθύνη στο Κοινοβούλιο. Για την απαλλαγή μιλώ, έτσι άλλο προπολογισμό που έχουμε κοινή ευθύνη, αλλά στην απαλλαγή δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να δεχθούμε να ε, ε, μας φέρεστε σαν να είμαστε απλώς μια αρχή που απευθύνει συστάσεις. Καθόλου συστάσεις. Είναι η αρχή που εγκρίνει και έχει τον τελευταίο λόγο το κοινοβούλιο. Πάρα πολύ σύντομα, Ναι. Σημειώνουμε ε, τη νομιμότητα του Κοινοβουλίου και ε, στο θέμα της απαλλαγής. Γι' αυτό κάνουμε και διάκριση ανάμεσα στο θέμα του προπολογισμού και της απαλλαγής και ξέρουμε ότι έχετε διακριτό ρόλο εκεί να διαδραματίσετε κι εσείς και θα τα αναφέρω αυτά στο Συμβούλιο και να είστε βέβαιοι ότι θα δώσουμε συνέχεια στη δήματά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, και στα Ισπανικά. Ο Υπουργός. Ευχαριστώ. Εξαντλήθηκε λοιπόν εδώ η συζήτηση για το σημείο 6 στην ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ Υπουργέ, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και ε, το Ελεγκτικό Συνέδριο για την παρουσία σας. Μην φύγετε κύριε Επίτροπε, ούτε το Ελεγκτικό Συνέδριο παρακαλώ, γιατί έχουμε και άλλο θέμα παριθμών 7 που σας αφορά. Και έχω πολύ ευχάριστα νέα για όλους σας κυρίες και κύριοι. Θα αναλάβει την Προεδρία αυτή τη στιγμή ο κύριος Μπάρτ Στάς που είναι πάντα ευχάριστα νέα. Ευχαριστώ πολύ Υπουργέ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 Καλησπέρα σα, συνάδελφοι. Ζητώ συγγνώμη που απουσίασα στην αρχή τη συνεδρίαση, αλλά είμαι σκιώδη εισηγητή και στην Επιτροπή Περιβάλλοντο και χρειάστηκε να είμαι εκεί. Και είναι και διαδικασία συναπόφαση για τα μεταλλαγμένα και βεβαίω έπρεπε να εκπροσωπήσω εκεί την ομάδα μου. Ερχόμαστε λοιπόν στο σημείο 7, απαλλαγή για το 2009 ε, σε έκθεση, έτσι, γενικός προπολογισμό της Ένωσης είναι αυτό. Ο συγητής μα είναι ο κύριο Χατζημαρκάκης. Γιώργο, μπορείς να κάνεις μια εισαγωγή στην έκθεσή σου και απευθύνομαι και στο ελεγκτικό συνέδριο αν θέλει να μιλήσει ευχαρίστω και ο Επίτροπος βεβαίω για να έχουμε μια πρώτη αντίδραση. Okay. Okay, that's good. Α, επιθυμεί το ελεκτικό συνέδριο να πάρει το λόγο μετά τον κύριο Χατζημαρκάκη. Ωραία. Πρώτο εισηγητή όμω και μετά να ζητάτε και το λόγο υπόλοιποι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ στα φλαμανδικά ο κύριο Χατζημαρκάκη. Κρίμα που έφυγε το Συμβούλιο βέβαια. Συνεχίζει στα αγγλικά ο μιλητή. Ορισμένα από τα θέματα ήδη όμω ετέθησαν. Αξίζει τον κόπο να σημειώσουμε ότι το Συμβούλιο με διπλή ιδιότητα και το τόνισε, είναι και θεσμικό όργανο και ως θεσμικό όργανο θέλει να δώσει απαλλαγή, αλλά η άλλη ιδιότητα που τείνουν να ξεχνούν είναι η εκτέλεση του προϋπολογισμού. Είναι η ιδιότητα του διαχειριστή των ταμείων και των γεωργικών δαπανών και των διαρθρωτικών ταμείων και των περιφερειακών στα κράτη-μέλη. Αυτή λοιπόν η δεύτερη ιδιότητα δεν λειτουργεί πάρα πολύ σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε την ευκαιρία να σας εισαγάγω στην ε, έκθεση για την απαλλαγή του 2009. Πριν μπούμε στην πολιτική ε, συζήτηση και στα πολιτικά ζητήματα, θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω τη δομή της έκθεσής μου. Μετά την εισαγωγή θα βρείτε πέντε κεφάλαια, A, B, C, D, E. Το κεφάλαιο Α αφορά ε, γενικά θέματα ε, που είναι και το κεφάλαιο ε, πρώτο του ελεγκτικού συνεδρίου. Το δεύτερο κεφάλαιο B είναι για τα ειδικά, όχι τα γενικά πλέον ευρήματα ε, του Συμβουλίου, του Ελεκτικού Συνεδρίου, συγγνώμη, σε ειδικού τομεί όπω είναι η παιδεία, η εξωτερική βοήθεια, η γεωργία, οικονομικά και χρηματοπιστωτικά κτλ. Και μετά Έχουμε ένα νέο κεφάλαιο, το κεφάλαιο Γ και Δ, C και D. σε περίπτωση που αναβάλουμε την απόφαση απαλλαγής. Αν υποστηριχθεί λοιπόν η αναβολή της απόφασης, το κεφάλαιο Γ αναφέρεται στους λόγους της πιθανής καθυστέρησης ή αναβολής απόφασης. Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει η Επιτροπή μας να καθορίσει ε, τα επόμενα βήματα που αναμένει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό είναι στο ΔΕΛΤΑ. Ανάληψη περαιτέρω δράσης και προς υποβολή έγγραφα. Σε περίπτωση που θα χορηγήσουμε την απαλλαγή, τα κεφάλαια Γ και Δ καθώς και αντίστοιχες τροπολογίες θα καταπέσουν και φτάνουμε στο κεφάλαιο Ε στις δράσεις προτεραιότητας. Και καταλαβαίνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζει τα κεφάλαια Γ και Δ να καταπέσουν και να μην παίξουν κανένα ρόλο. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε όλα αυτά τα κεφάλαια και αυτό σας εξηγώ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο, τον κύριο Σεμετά, γιατί ήταν υπερδραστήριος ε, στην όλη διαδικασία. Μας βοήθησε να βρούμε απαντήσεις για την επόμενη τη μελλοντική δηλαδή πολιτική στρατηγική, γιατί περί αυτού πρόκειται στην έκθεση, τι να κάνουμε στο μέλλον. Επανειλημμένα έχουμε πει ότι επί 16 συναπτά έτη είναι ανετική η δήλωση αξιοπιστίας. Και ήδη από την εποχή ε, της Επιτροπής Μπαρόσο 1 ε, είχαμε στρατηγικό στόχο για θετική δήλωση αξιοπιστίας, πράγμα που δεν επετεύχθη. Μετά, θα βρείτε και κάποιους ισχυρισμούς ε, στα κεφάλαια αυτά και χαίρομαι πάρα πολύ που ο Επίτροπος άρχισε από την πρώτη μέρα των συζητήσεών μας να μας δίνει στοιχεία αυτά τα αιτήματά μας και συνεχίζεται η συνεργασία μας, συνεχίστηκε σε εβδομαδία βάση, διότι βεβαίως ο στόχος είναι πάντα οι βελτιώσεις, αλλά για να γίνει αυτό ε, χρειάζεται πρώτα αποτελέσματα. Να σας πω τα σημαντικότερα στοιχεία σε έξι βήματα. Πρώτον, κάτι που μόλις συζητήσαμε και προηγουμένως και με την Προεδρία του Συμβουλίου και αυτό είναι το θέμα των εθνικών ε, δηλώσεων διαχείρισης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό είναι και παραμένει ένα πολύ σημαντικό ε, σημείο στα αιτήματα του Κοινοβουλίου. Εθνικές ε, λοιπόν δηλώσεις με υπογραφή του εκάστοτε Υπουργού Οικονομικών. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί κάτι τέτοιο από πλευράς πολιτικής. Θα μπορούσαμε όμως να ε, το επιτύχουμε σε ένα πρώτο βήμα, επαναλαμβάνω πρώτο βήμα σε επίπεδο διοικητικό, διαχείρισης. Και συγχαρητήρια κύριε Σεμετά και σας ευχαριστώ γιατί έχετε φέρει ένα κατάλογο με σαφή κριτήρια. Και διαβιβάστε και αυτό σε όλα τα μέλη της Επιτροπής μας σήμερα το πρωί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας φέρατε από μόνο σας αυτό τον κατάλογο σαφών κριτηρίων. Περιμένετε από τα κράτη-μέλη να κάνουν αυτά για τη ε, δήλωσή τους σε επίπεδο διαχειριστικό πλέον και όχι πολιτικό για το πώς εκτελούν τον κοινοτικό προπολογισμό. Επίσης είχατε την καλοσύνη να αρχίσετε με ένα κατάλογο που κατονομάζει τέσσερα κράτη-μέλη που κάτι δίνουν, κάποια δήλωση αξιοπιστία, ε, υπόλοιπα πάρα πολύ λιγότερα, αλλά είχατε την καλοσύνη να μας δώσετε και εκεί κάποια στοιχεία για το που πορευόμαστε και πώς ε, ανταποκρίνονται στα κριτήρια που έχετε βάλει εσείς στα κράτη αυτά και θα ήθελα να σας καλέσω βεβαίως να συνεχίσετε να πιέζετε και τα άλλα κράτη-μέλη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά ένα πρώτο βήμα και μόνο. Και επίσης θα θέλαμε να το εφαρμόσετε, να το ε, προωθήσετε αυτό στο μέλλον και στον επόμενο δημοσιονομικό κανονισμό και στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ένα δεύτερο θέμα τώρα αφορούσε τη μεγαλύτερη ε, λογοδοσία των επιτρόπων ή της Επιτροπής ως συλλογικό σώμα. Όταν εγκρίνεται η συνθετική έκθεση ή η ετήσια έκθεση πεπραγμένα. Ε, ζητώ συγγνώμη από τον Επίτροπο Χάν καταρχάς. Όταν βλέπουμε τα αποτελέσματα της επιτροπης ως συλλογικο σωμα οταν εγκρινεται η συνθετικη εκθεση η η αιτησια εκθεση πεπραγμενα δράσης, έκθεση πεπραγμένου. Ο Επίτροπος λέει ότι δεν ήξερε τη διατύπωση, αλλά ήξερε τις αρχές και μόνο. Εντάξει, το σημειώνουμε. Παρ' όλα αυτά, είναι σαφές ότι χρειάζεται μεγαλύτερη λογοδοσία των ίδιων των Επιτρόπων για τα πεπραγμένα τους, γιατί φέρουν και τελικά πολιτική ευθύνη, έτσι δεν είναι. Και καλωσορίζω πάρα πολύ το γεγονός ότι το θέμα αυτό ετέθη από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον ίδιο ε, στο Σώμα των Επιτρόπων. Και κυκλοφόρησε και ένα ιστορικό σημείωμα όπου ε, αναφέρεται ότι στο μέλλον θα πρέπει οι γενικοί διευθυντές να ενημερώνουν τους επιτρόπους τους για τα προβλήματα, για τις επιφύλαξεις, τουλάχιστον άπαξ ετησίω. Πλην όμως θέλουμε και στη συνθετική σας έκθεση να τα αναφέρετε αυτά και με την εξή μορφή. Μια εκτίμηση ή αξιολόγηση για τις επιδόσεις των κρατών μελών, αν τα πηγαίνουν καλά ή αν δεν τα πηγαίνουν καλά. Είχαμε ε, συζητήσει αυτό το θέμα τον κύριο Σεμετά και νομίζω αυτή η συνθετική έκθεση είναι σκόπιμο να περιλαμβάνει ένα πίνακα επιδόσεων ή δεν ξέρω κάποια εκτίμηση εν πάση περιπτώσει για το πώς ε, εκτελούν τον προπολογισμό τα κράτη-μέλη. Επόμενο θέμα. Διακοπή και ε, αναστολή πληρωμών. Η διακοπή πληρωμών των κοινοτικών ε, κονδυλίων είναι νέο στοιχείο που εισήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί πάρα πολύ ειλικρινά και πάρα, με πολύ μεγάλη διαφάνεια το 2010 εκδώσατε και ένα κατάλογο των διακοπών πληρωμών. Είναι μια διαδικασία εν εξελίξη το είπα και προηγουμένω όταν ήρθε ο κύριο Μπέκτσάι, ο Υπουργό. Όλα τα προγράμματα στην Αγγλία, για παράδειγμα, έχουν διακοπεί και έχουν εξαιρεθεί από τον κατάλογο. Σα ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ για τη διαφάνεια αυτή. Και δεδομένου ότι είναι νέο αυτό το μέσο, ανάγεται μόλις το 2009, είναι δύσκολο να έχει κανείς στοιχεία από προηγούμενες εποχές. Αλλά υπήρξαν και άρσεις μάλλον ε, αναστολές πληρωμών για πολιτικούς λόγους. Και θα θέλαμε να μας δώσετε και αυτό τον κατάλογο και δεσμευτήκατε άλλωστε ο ίδιος να το πράξετε. Είναι πολύ σημαντικό. Παρ' όλα αυτά, χρειάζεται κάποιος αυτοματισμός. <coughs> Δηλαδή πότε διακόπτονται κάποιες πληρωμές ή αναστέλλονται αργότερα. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τον κατάλογο που μας δώσετε ήδη με σαφή κριτήρια τα οποία θα οδηγούν σε διακοπή πληρωμών. Θα ήθελα να σας θυμίσω όμως ότι στον κανονισμό του Συμβουλίου υπάρχει ακόμα ε, όρος δίνανται. Είναι ακόμα δυνητική η διάταξη. Ακόμα και αν είναι δυνητική η διάταξη θα πρέπει να προβλέπουμε ε, και διακοπή χωρίς πολιτική παρέμβαση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εδώ και το μεγαλύτερο εμπόδιο θέλετε είναι η ανάκτηση των πόρων. Ε, το υπενήχθη και ο Υπουργό. Εσεί έχετε δεσμευτεί, κύριε Επιτροπέ, σε μια επιστολή που μα απευθύνεται να μα στείλετε ένα μνημόνιο, ε, ένα memorandum, με ε, μια επισκόπηση όλων των, ε, χρημα... των οικονομικών διορθώσεων του παρελθόντος και επίση θα θέλαμε να σας ζητήσουμε ε, να μας πείτε πόσα χρήματα έχουν επανιστρέψει στα ταμεία σας. Ε, τα, ποσά. Φαντάζομαι θα είναι χαμηλό το, το, πραγματικό ποσό. Και μπορεί αυτό να σημαίνει ότι ο φορολογούμενος πληρώνει δύο φορές. Λοιπόν, σας παρακαλώ δώστε μας αυτά τα στοιχεία και θα τα ξανασυζητήσουμε. Και μας έχετε υποσχεθεί ότι θα το κάνετε μέχρι τον Απρίλιο. Επόμενο θέμα ή εκθέσει αξιολόγησης, ε, οι μελλοντικέ. Αυτό ε, αφορά το άρθρο 318 της συνθήκη. Για πρώτη φορά το 2011, για το έτος 2010 θα κατατεθεί τέτοια έκθεση. Χαιρόμαστε που δεσμεύεστε να φέρετε και πάλι βασικά κριτήρια. Δεν μιλήσατε για τους βασικούς δείκτες επιδόσεων, αυτό που θέλω εγώ είναι να έχουμε αιτήσια συζήτηση ε, για ε, οικονομικό έλεγχο των επιδόσεων. Πώς ελέγχουμε δηλαδή την αποτελεσματικότητα του αν πιάνουν τόπο τα χρήματα. Δεν απαντήσατε, ε, φαντάζομαι ότι θα απαντήσετε. Αν θα ορίσετε και ειδικό πρόσωπο για αυτή την έκθεση επιδόσεων. Και θα θέλαμε να καλέσουμε το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο να παίξει πιο αποφασιστικό ρόλο εκεί. Ε, στην αξιολόγηση των επιδόσεών σας και των δικό σας δηλαδή σε σχέση με την έκθεση αυτή και να συμμετέχει στην ετήσια συζήτηση που θα θέλαμε να σας καλούμε να έχουμε για τη δική σας πλέον επίδοση. Ένα τελευταίο θέμα έχει να κάνει με την απλούστευση. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήδη δεσμευτήκατε και πάλι, κύριε Επίτροπε, να εκδώσετε κατευθυντήριες γραμμές για την απλούστευση. Γνωρίζω ότι ε, το πλαίσιο είναι δημοσιονομική δημοσιονομικοί κανονισμοί γι' αυτό και η πρόταση θα γίνει τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Μέχρι τότε όμως θα θέλαμε να σας δώσουμε απαλλαγή. Οπότε και εσεί θα θέλατε, θα θέλαμε εκ των προτέρων να μας δώσετε αν όχι κατευθυντήριες γραμμές, κάποια πρακτικά παραδείγματα. Πού θέλετε, πού πιστεύετε ε, να εφαρμόσετε αυτές τις απλουστεύσει. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι διαπραγματεύσει, και έχω τη χαρά να σας ενημερώσω γι' αυτό με τον Επίτροπο τον κύριο Σεμετά και ε, το ιδιαίτερο γραφείο του και τι υπηρεσίε του είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο προχωρούμε πολύ καλά. Ε, δεν μας έχουν ικανοποιήσει σε όλα τα σημεία, δεν μας έχουν απαντήσει. Μπορεί να γίνει αυτό, το δείτε και στην επιστολή που σας διαβιβάστηκε. Ε, πάντως είμαι πεπισμένος ότι όχι μόνο σε καλό δρόμο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά μέχρι τέλη Μαρτίου και πριν ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή μας σε βάση περιπτώσει, θα έχει απαντήσει σε όλα τα σημεία. Για το λόγο αυτό έχω αφήσει ανοιχτό το θέμα αν θα δώσουμε ή όχι την απαλλαγή. Αυτά. Και ήταν αυτό ένα τρόπο να καλωσορίσω και να χαιρετήσω την πολύ καλή αρχή των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, έχουμε ακόμα την ευκαιρία ή τη δυνατότητα να το αλλάξουμε. Οπότε, θέλω να σας πω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, αλλά είμαστε μόνο στα μισά του δρόμου. Έχουμε άλλο τόσο να διανύσουμε. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σεγητά. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο που μας έστειλε αυτή την επιστολή. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη και πάρα πολύ διαφωτιστική. Θα ήθελα να δώσω πρώτα την ευκαιρία στο ελεγκτικό συνέδριο να απαντήσει. Η κυρία Καλγιολέιτ. αν ε, προφέρω σωστά το όνομά σας, θέλετε πρώτα εσείς να απαντήσετε, να αντιδράσετε στα όσα είπε ο κύριος Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα και πάλι το ελεγκτικό συνέδριο δεν θέλει να αναμειχθεί σε πολιτική συζήτηση σχετικά με την απαλλαγή. Δεν είναι αυτή αυτός η αρμοδιότητά μας, αλλά χαιρόμεθα μπορούμε να συμβάλλουμε στην συζήτηση. Δεν έχουμε βασικά θέματα για το πώς ε, ε, το, αν το ψήφισμα περί απαλλαγής αντιπροσωπεύει ε, τις διαπιστώσεις μας από τον έλεγχο και ε, είμαστε ευγνώμονες στον εισηγητή για αυτήν την ενδελεχή συζήτηση που είχαμε για όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στον κύριο Σεμετά. Δύο έχουν ζητήσει, ο κύριος Φιέλνερ και η κυρία Ιβάνοβα προς το παρόν από συναδέλφους. Κανείς άλλος συνάδελφος δεν θέλει το λόγο. Όχι, καλώς. Ο Επίτροπος τότε έχει την ευκαιρία να απαντήσει, να υπερασπιστεί την υπόθεσή του και να απαντήσει στις συμπληρωματικές ερωτήσεις του κυρίου Χατζημαρκάκη. Ευχαριστώ. Κύριος Επίτροπος, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε συγητά, αξιότιμα Μαμέλη από την παρουσίαση της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου τον Νοέμβριο 2010. Ένας διάλογος ενδελεχής και καρποφόρος έλαβε χώρα ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή. Περιλαμβάνονται ορισμένα θέματα και αιτήματα στα οποία η Επιτροπή θα απαντήσει λεπτομερώς. Για τη σημερινή μας συζήτηση θα ήθελα να επικεντρωθώ πάνω στις απαντήσεις στα έξι θέματα της παραγράφου 113 του σχεδίου έκθεσης και που αναφέρονται στην επιστολή που έστειλα την τελευταία πέμπτη, την περασμένη πέμπτη στον πρόεδρο και στον εισηγητή πρόκειται για τις υποχρεωτικές δηλώσεις της εθνικές διαχείρισης Έχετε όλοι αυτό το αίτημα εδώ, την, ε, την πρόταση. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι σε αυτό το στάδιο οι εθνικές δηλώσεις δεν παρέχουν ή παρέχουν μόνο εν μέρη τις πληροφορίες που απαιτούνται ε, για την διαδικασία δήλωσης αξιοπιστίας επιτροπής. Επίσης υπάρχει τεχνη, ε, τεχνική κατευθυντήρια γραμμή για τις δημόσιες αρχές για το πώς ε, να προσθέσουν αξία σε αυτές ε, για τις δηλώσεις αξιοπιστίας. Αναφέρονται σε βασικά στοιχεία ε, της πρότασης ε, για την αναθεώρηση ούτω ώστε τα αξιοσοδοτημένα σώματα να μπορούν να καταρτήσουν μια ετήσια εθνική δήλωση ε, που να βασίζεται σε λεπτομερή έκθεση και να ακολουθεί ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο. Θα ήθελα να σας ζητήσω να υποστηρίξετε αυτό το νέο λογιστικό μέσο που είναι σύμφωνο με τον κανονισμό με αυτό το, τη νέα, η νέα διαδικασία αυτή θα αξιολογηθεί πάνω σε αυτήν την βάση η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα ασκήσουν πίεση στα κράτη-μέλη ούτως ώστε να λάβουν σοβαρά υπόψη αυτό, αυτό το νέο μέσο λογοδοσίας. Το δεύτερο θέμα αναφέρεται στη δομή διακυβέρνησης της Επιτροπής, ε, κυρίως ε, την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων ε, του Αρμοδίου Επιτρόπου και των Διευθυντών. Ο εισηγητής ανέφερε στο σχέδιο έκθεσης ότι αυτή η έκθεση θα έπρεπε να υπογραφεί σε πολιτικό επίπεδο, δηλαδή να συνυπογραφεί από τον Αρμόδιο Επίτροπο και από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Συγκεφαλαιωτικής Έκθεσης. Η Επιτροπή βασίζει την διαδικασία για την αξιοπιστία σε καθαρό διαχωρισμό ανάμεσα στο διοικητικό επίπεδο και στο πολιτικό επίπεδο. Ο Γενικός ε, Διευθυντής υπογράφει την δήλωση και το Σώμα των Επιτρόπων ε, υιοθετεί ε, συλλογικά την συγκεφαλαιοτική έκθεση. Ωστόσο, συμφωνώ ότι, ότι και τα δύο υποστηρίζουν δύο πυλώνες στο ίδιο οικοδόμημα. Γι' αυτό ζήτησα από τις εσωτερικές υπηρεσίες να ενημερώσουν τις οδηγίες. Ο Γενικός Διευθυντής θα διευκρινίζει ότι έχει πλήρως ενημερώσει τον Επίτροπο για τα βασικά θέματα και κυρίως για τις επιφυλάξεις που λαμβάνονται υπόψη στην, στην έκθεση δραστηριοτήτων. Αυτές οι οδηγίες έχουν δημοσιοποιηθεί και γνωστοποιηθεί στις υπηρεσίες και ο πρόεδρος και εγώ επιμείναμε στην τελευταία συνεδρίαση του Σώματος για την σημασία αυτών των πληροφοριών για τον κάθε έναν από αυτούς και για το Σώμα των Επιτρόπων στο σύνολό του και θα γνωστοποιηθούν στα επίσημα πρακτικά της Επιτροπής και θα αποσταλούν επίσης αυτή την Επιτροπή. Το τρίτο θέμα αναφέρεται στην καθιέρωση της αυτόματης διακοπής και αυτόματης αναστολής των πληρωμών μόλις υπάρχει σημαντική ανεπάρκεια στην λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου. Για την περίοδο μέχρι το 2013 έχουμε μια σαφή νομική βάση για την αναστολή και την διακοπή. Και η Επιτροπή χρησιμοποιεί αυτό το μέσο όπως αποδείχθηκε από τον κατάλογο όλων των, ε, των διαστηριοτήτων διακοπής και αναστολής το 2010. 15 απαιτήσει που έχουν καθιερωθεί σε συνεργασία με το ελεγκτικό συνέδριο χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής για να αξιολογήσουν ε, τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου ε, των κρατών και την ε, πολιτική συνοχή. Οι οδηγίες για την προετοιμασία της ετήσιας έκθεσης έχουν συμπληρωθεί με νέες υποχρεώσεις για την παροχή λεπτομερέστερων πληροφοριών για τις αποφάσεις είτε διακοπής είτε αναστολής των πληρωμών και συζητήσαμε σήμερα για ακόμα περαιτέρω βήματα σε αυτόν τον τομέα ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο αυτοματισμό και για να συζητήσουμε με τις υπηρεσίες τι περαιτέρω μέσα ε, και πρωτοβουλίες θα μπορούσαμε να αναλάβουμε σε αυτόν τον τομέα. Το τέταρτο θέμα είναι οι διορθωτικοί μηχανισμοί και η Επιτροπή δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει με τον εισηγητή ότι η καλή τήρηση των κανόνων έχει πρωτεύουσα σημασία για την προστασία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πολιτική συνοχή πρέπει να καλύπτουν όλα, όλες τις, τα πλήρωτα ποσά τα κράτη-μέλη αλλά και χρειάζεται ανάκτηση από τον τελικό δικαιούχο. Συνεπώς, η καθιέρωση ενός συστήματος ανάκτησης ε, αποτελεί μέρος της υποχρεωτικής επαλήθευσης και ελέγχου στην αρχή της περίοδου προγραμματισμού. Ε, τώρα, ε, μετά την εφαρμογή των συστημάτων υπόκειται σε αξιολόγηση τακτική και θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην, στην απόδοση των κρατών μελών, στα αποτελέσματα των κρατών μελών ως προς την ανάκτηση. Είχαμε πολλές συνεδριάσεις με εθνικές αρχές ούτως ώστε να αναπτύξουμε ένα σύστημα ούτως ώστε να διορθωθούν τα πιο επικίνδυνα συστήματα ούτως ώστε να έχουμε καλή ανάκτηση. Αυτές οι δραστηριότητες θα συνοψιστούν σε ένα μνημόνιο το οποίο θα αποστείλω στο Κοινοβούλιο πριν από το τέλος του μηνός Απριλίου. Θα ήθελα τώρα να περάσω στο πέμπτο θέμα που ανέφερε ο εισηγητής και που αναφέρεται στον αξιολογητή επίδοσης που εισάγεται από το άρθρο 318 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Αυτό το νέο μέσο αναφοράς θα μας δώσει μια καλή ευκαιρία για να βελτιώσουμε περαιτέρω την αξιολόγηση της επίδοσης και της προστιθέμενης αξίας των προγραμμάτων και πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιώντας δείκτες. Θα παρουσιάσει η Επιτροπή πριν από το τέλος του Μαρτίου σε γενικές γραμμές ένα κείμενο που θα βασίζεται στο άρθρο 318 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο έκτο και τελευταίο θέμα του σχεδίου έκθεσης, ο εισηγητής ζητά την καθιέρωση μιας νέας λογικής δαπανών που θα στοχεύει μεταξύ άλλων στη βελτίωση της ποιότητας των δαπανών για να εξασφαλίσει ρεαλιστικές δαπάνες. Όπως γνωρίζετε, η απλούστευση είναι μια υποχρέωση βασική που επανέλαβε πολλές φορές ε, η Επιτροπή, κυρίως στην ανακοίνωση για την ε, επισκόπηση του προϋπολογισμού και επίσης στην επισκόπηση του δημοσιονομικού κανονισμού. Η απλούστευση θα είναι σημαντικό μέρος της εργασίας μας για την προετοιμασία και διαπραγμάτευση των μελλοντικών προγραμμάτων. Η Επιτροπή ήδη εργάζεται για διάφορες επιλογές για να απλουστευτούν οι κανόνες, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή όλων των πρωταγωνιστών και εμπλεκομένων στην επόμενη γενεά προγραμμάτων. Αυτό το συζητήσαμε και ε, καταρτήσαμε κατευθυντήριες γραμμές για την απλοποίηση των υπηρεσιών της εργασίας των υπηρεσιών όταν θα προετοιμαστεί η νομοθεσία για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Θα υπάρξει μια συνεκτική προσέγγιση για την μελλοντική απλούστευση. Ε, Πρωτού κλείσω θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η ανάλυση μας ήδη δείχνει ότι ένας περιορισμένος αριθμός κρατών μελών δίνει, ε, ε, έχει λάβει υπόψη της επιφυλάξης του Γενικού Διευθυντή και ένα σημαντικός αριθμός διακοπών και αναστολών ε, και δημοσιονομικών διορθώσεων έχουν γίνει. Πρέπει να εξαγάγουμε συμπεράσματα από το γεγονός αυτό και να συγκεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στις ασθενέστερες αρχές με ενισχυμένη βοήθεια και όπου αυτό απαιτείται με προληπτικά μέτρα, δηλαδή αναστολή, διακοπή πληρωμών και διορθωτική και αλλού με διορθωτικά μέτρα και με μέτρα κλεισίματος και αυτό θα το πράξει η Επιτροπή. Συνεπώς σας παρουσίασα τις συγκεκριμένες πράξεις και μέτρα τα οποία η Επιτροπή έχει, έχει αναλάβει αναλάβει ως απάντηση στις ανησυχίες που εκφράζονται στην έκθεση και αυτό θα σας βοηθήσει να λάβετε τις καλές αποφάσεις εφόσον υπάρχουν δύο σενάρια επιτάπητος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστούμε για τις απαντήσεις σας. Νομίζω ότι ε, μπορώ και εγώ να καταθέσω τη μαρτυρία μου ότι ήταν πάρα πολύ εντατική αυτή η άσκηση. Έχουμε ζήσει ε, τώρα αρκετές ε, τέτοιες απαλλαγές όπου η ανταλλαγή ε, απόψεων ήταν πάρα πολύ εντατική μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εισηγητού και όχι μόνο επίτροπος σε μετά αλλά και άλλοι επίτροποι και πολλοί ε, είχαν ε, την ευκαιρία προσωπικά να συζητήσουν ε, κάτι κατηδία με τον ε, εισηγητή και χαιρόμαστε και σας ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Πιέλνερ, μετά η κυρία Ιβάνοβα και μετά εσείς να κλείσετε κύριε εισηγητά. Ευχαριστώ πολύ. Πριν από έξι χρόνια, νέος ευρωβουλευτής, θυμάμαι ότι δεν μου άρεσε πώς μιλάει κανείς όταν παίρνει το λόγο. Δεν ξέρω τι εξαιρετικός που ήταν ο εισηγητής, τι ωραία πράγματα που έκανε, η Κομισιόν κλπ και μετά ξεδεύουν τον υπόλοιπο χρόνο τους. Ναι, αλλά διαφωνώ σχεδόν με τα πάντα. Και υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει ακριβώς το ίδιο και με μένα. Δεν ξέρω αν άλλαξα στα έξι αυτά χρόνια που είμαι ευρωβουλευτής. Θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντας τον κύριο Χαζημαρκά για τη δουλειά του, για αυτά που μας είπε. Σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ και ευχαριστώ και την Κομισιόν. Γιατί είχαμε πολύ γόνιμη συνεργασία. Είναι πολύ ωραίο η διαδικασία απαλλαγή ε, να δούμε πριν καν την ψηφίσουμε πόσο ωραία κινήθηκε. Δηλαδή θέσαμε ερωτήματα, υπογραμμίσαμε ορισμένα σημεία, δημιουργήθηκε ένα δυναμικό αλλαγή που την χρειάζεται η Κομισιόν. Ωστόσο, και εδώ αρχίζουμε τις ενστάσεις, το υπόλοιπο της ομιλίας μου. Δυστυχώς θα, είμαι κάπως, ε, θα μιλήσω κάπως περισσότερο από εδώ και μπρος. Θα μείνω κι εγώ στο σημείο Δέλτα. Μπορούμε να συζητήσουμε κι άλλο το τι θέλουμε, τι έγραφα, τι δράσεις, αν υπάρχουν επαρκή επιχειρήματα για αναβολή ή όχι. Αλλά ας ξεκινήσουμε βλέποντας την ουσία. Την ουσία. Αυτόν που μας λέει ο εισηγητής. Πρώτον για τις εθνικές δηλώσεις διαχείρισης. Το έχουμε συζητήσει αρκετά και συμφωνούμε. Είναι κάπως περίεργο να πούμε ότι αυτό το θέλουμε από την Κομισιόν. Ουσιαστικά από τις κυβερνήσεις το θέλουμε. Αλλά πρέπει να πούμε ότι η Κομισιόν και αυτή μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω και ευχαριστώ πολύ τον ε, Επίτροπο για το έγγραφο που μας έστειλε όπου λέει ναι δεχόμαστε να κάνουμε κάτι παραπάνω υπάρχει ακόμα περιθώριο και άλλο περιθώριο βελτίωσης. Ναι μεν χρειάζεται να το συζητήσουμε κι άλλο μεταξύ μας τι προκλήσεις υπάρχουν σχετικά με τις εθνικές αυτές δηλώσεις διαχείρισης Έχουμε κράτη που είναι ομοσπονδιακής δομής, έχουμε πρόβλημα προθεσμιών, πόσους χρόνους δηλαδή απαιτείται προκειμένου το εργαλείο αυτό να αποδώσει και τέλος φυσικά είναι και το θέμα της υπογραφής των υπογραφών. Μακάρι στη Σουηδία ο υπουργός Οικονομικών να μπορούσε να υπογράψει αλλά δεν θα ήθελα να είναι κάτι που να είναι μόνο συμβολικής αξίας, να είναι ουσία, πραγματικά να επηρεάζει την ουσία, την ποιότητα. Και στο σημείο αυτό έρχεται η Κομισιόν και μας μιλάει για ορισμούς, μας μιλάει για την ουσία, πώς να λειτουργεί το σύστημα και να μην επιμένουμε υπερβολικά στο, στην υπογραφή. Δεύτερον, εκθέσεις δραστηριοτήτων. Ναι, να υπογράφει τις εθνικές δηλώσεις ο υπουργό Οικονομικών, αλλά εξίσου λογικό είναι και ο Επίτροπος να υπογράφει την ε, έκθεση δραστηριότητας. Βέβαια, αυτό αυξάνει τον, την ευθύνη που έχει ο καθένας. Οι γενικοί διευθυντές Φερρυπίν θα πρέπει και αυτοί να έχουν ευθύνη και νομίζω ότι εδώ συμφωνούμε με την θέση που λέει ότι οι εκθέσεις δραστηριότητας θα πρέπει να μετράνε περισσότερο. Να το χρησιμοποιεί η Επιτροπή στο συλλογικό σώμα και μεταξύ των γενικών διευθυντών και με τον, σε σχέση με τον Επίτροπο να μην είναι συμβολικό μόνο το θέμα, να έχει και πρακτική αξία. Το τρίτο σημείο Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο εισηγητής μας και είναι ζωτική σημασία το γάμα. Μπορούμε να συζητήσουμε αν θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό ή λιγότερο υποχρεωτικό. Το σημαντικό για μένα είναι να ξέρουμε πότε η Κομισιόν διακόπτει μια δράση και αν δεν διακόψει να τους πούμε γιατί δεν εφαρμόζετε τους κανόνες, αν υπάρχει περιθώριο ελιγμών καλώς. Αρκεί να δούμε πώς το χρησιμοποίησαν. Πρέπει η Επιτροπή να έχει την ευθύνη στο θέμα αυτό. Το ΔΕΛΤΑ για τις διορθώσεις είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Το ε λατινικό είναι επίσης σημαντικό για το νέο σύστημα του 318 Βέβαια μου είναι δύσκολο να υπολογίσω ποια θα είναι η τελική διαφορά. Ίσως επειδή είμαστε ακόμα στην πρώτη φάση εφαρμογής. Πάντως είναι και αυτό ένα ερώτημα. Το τελευταίο σημείο, το λατινικό F, είναι δύσκολο να είναι κανείς εναντίον μιας νέας λογικής για τις δαπάνες. Χρειάζεται όμως έλεγχος. Ναι, να έχουμε ένα νέο σύστημα δαπανών Αλλά πάλι θα πρέπει να δούμε την ουσία της εφαρμογής. Είναι εφαρμόσιμο ή όχι. Στο ΕΛΚ το συζητήσαμε ήδη το θέμα και ξέρω ότι υπάρχουν συνάδελφοι που θα θέσουν ε, ερωτήματα σχετικά με το προσωπικό, Φερρυπίν. Αυτό δεν είναι στο, στο ΔΕΛΤΑ, στο οποίο αναφέρθηκα πριν. Θα επανέλθω σε αυτό όμως. Ή θα επανέλθουμε μάλλον σε αυτό και σε ορισμένα άλλα σημεία πειθαρχικών ε, διώξεων, ε, δράσεων της ε, Κομισιόν. Θα πρέπει όλα αυτά να τα ξαναδούμε. Να ξαναδούμε πάλι την επιστολή και τις προθέσεις που υπάρχουν στην επιστολή αυτή της Κομισιόν έτσι ώστε να μετράει, να βαρύνει αυτή η διαδικασία απαλλαγή. Και είμαι σίγουρος ότι θα συνεργαστούμε και με τον εισηγητή και με την Κομισιόν. Πάντως σε μεγάλο βαθμό συμφωνούμε με τα βασικά σημεία. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Νομίζω η παρέμβασή σας ήταν αρκετά μετριοπαθής. Η κυρία Ιβανόβα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν και εγώ ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πάρα πολύ σοβαρή δουλειά του κύριε Χατζημαρκάκη. Επίσης ευχαριστώ και τον Επίτροπο που ήρθε και έχει έρθει και στις ακροάσεις και μας βοήθησε να επισημάνουμε τα ασθενή σημεία στην εκτέλεση του προπολογισμού και ευχαριστώ και τον τύπο, τα μέσα ενημέρωσης που συχνά έχει κρούσει τον κόδωνο του κινδύνου για ασφάλματα, για παρατυπίες και μας βοηθάνε να βελτιώσουμε το σύστημα. Γενικά τα περισσότερα υπόθηκαν. Ο Κρίστεφερ κάλυψε τις απόψεις του ΕΛΚ στα επιμέρους σημεία. Δεν θα τα επαναλάβω λοιπόν κι εγώ. Συμφωνώ με τα επικριτικά σχόλια και την γραμμή πλεύσης του εισηγητή μας. Ιδιαίτερα επισημαίνω την πρόοδο που σημειώθηκε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό το μαρτυρεί και η έκθεση του συνεδρίου και αυτά που μας είπε η Επιτροπή. Θετικές επίσης οι προσπάθειες του Επιτρόπου των τελευταίων ημερών προκειμένου να μας παρουσιάσει τη θέση του ως απάντηση στην θέση του Κοινοβουλίου. Στη συνοχή έχουμε ένα υπέρβαση 5% αλλά ταυτόχρονα έχουμε μείωση διαχρονικά στα έξι σημεία που αναφέρθηκαν ε, σκοπεύω να υποβάλω μερικέ τροπολογίες στην έκθεση. Το πρώτο, η ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων ελέγχου. Συμφωνώ με την πρόταση του εισηγητή για να τονωθεί αυτή η διαδικασία με ορισμένα πρόστιμα. Προσθέτω ότι χρειάζομαστε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες και στοιχεία από την Κομισιόν για τους ποιοτικού ελέγχους κατά κράτος και κατά τομέα πολιτικής για να μπορούμε να αξιολογήσουμε, να συγκρίνουμε πώς ε, λειτουργούν αυτοί οι μηχανισμοί γιατί μικρό επίπεδο απάτης μπορεί να σημαίνει ότι το σύστημα ελέγχου να μην είναι επαρκές. Περισσότερα σφάλματα μπορεί να σημαίνει ότι το σύστημα ελέγχου αποδίδει περισσότερο. Δεν πρέπει αυτόματα να δακτυλοδειχτούμε κυβερνήσεις χωρίς να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Δεύτερο στοιχείο που μου παραξενεύει κάπως, με βάση την προφορική έκθεση δραστηριοτήτων του 2010 σε σχέση με το 2009, βλέπουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις τα διαφορετικά ταμεία οι απάτες οργανώνονται, προγραμματίζονται εκ των προτέρων. Οργανώνονται. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Πρέπει να το προσέξουμε. Να δημιουργούνται τέτοιες ευκαιρίες. Να το ελέγχουν αυτό και οι κυβερνήσεις και οι κομισιόν. Και τρίτο και τελευταίο, το χρονοδιάγραμμα της απαλλαγής και η επιτάχυνσή του. Πώς να εξηγήσω εγώ στις εκλογείς μου ότι σήμερα το 2011 συζητάμε την απαλλαγή του 2009. Πρέπει να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία θα γίνει πιο διαφανής, θα βλέπουμε τα ασθενή σημεία πιο γρήγορα, θα φροντίζουμε να διορθώνονται. Ο καθένας ανάλογα με τις ευθύνες του. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Ιβάνοβα. Έχει ζητήσει ο κύριος Γερμπράντη το λόγο πλέον. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και ο συνάδελφος Φιέλνερ μόλις έφυγε. Με ενέπνευσαν όμως τα λόγια του ότι είναι εδώ έξι χρόνια και σιγά σιγά έχει υιοθετήσει κάποια ήθη που κυκλοφώνουν στο κοινοβούλιο. Εγώ είμαι βουλευτή λιγότερο χρόνο, αλλά με ενέπνευσαν πραγματικά αυτά που άκουσα. Α μην γελιόμαστε. Έχουμε κάποια στοιχεία για την εκτέλεση του κοινοτικού προπολογισμού. Δεν υπάρχει κράτος μέλος και δεν υπάρχει ευρωβουλευτή που να έπρεπε να δώσει την απαλλαγή με αυτά τα στοιχεία. Εντάξει, στο παρελθόν ήταν πολύ χειρότερα και υπάρχουν βελτιώσεις αργά αλλά σταθερά και σιγά σιγά έχουμε μπει σε αυτή τη συνήθεια και σε αυτό ε, το να δεχόμαστε τα κακά στοιχεία και στο τέλος να δίνουμε την απαλλαγή. Ας μην γελιόμαστε, παραμένουν τρομακτικά τα στοιχεία, δεν θα πρέπει να χορηγήσουμε απαλλαγή. Εγώ δεν θέλω να προσαρμοστώ στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε εδώ προσπαθώ να παραμείνω σε ένα επίπεδο ε, ριζοσπαστικότητας, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η λέξη, ριζοσπαστισμού. Ε, πάντως αναρωτιέμαι, χρειαζόμαστε αυτά τα μικρά βήματα για να ε, βελτιώσουμε σιγά σιγά τα ποσοστά ή μήπως να δούμε κατάματα την πραγματικότητα και να είμαστε πιο ειλικρινείς ο ένας απέναντι στον άλλον ότι χρειάζονται πιο ριζοσπαστικά βήματα θαραλέα ε, για να κοιτάμε κατάματα τους εκλογής μας. Κανένας δεν πρόκειται κανονικά να δεχτεί να δώσει απαλλαγή. Δεν θα έπρεπε με αυτά τα στοιχεία. Πρέπει να σας πω ότι είχα τις ίδιες ερωτήσεις και κατά τη διάρκεια της ακρόασής σας κύριε Επίτροπε πριν από 1,5 χρόνο εθνικές δηλώσεις δεν θα πρέπει να είναι πιο ακραίες, δεν θα πρέπει να αναγκάσουμε τα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα τώρα που έχουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας και τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν περισσότερες ευθύνες. Ο υφυπουργό οικονομικών κρύφτηκε πίσω από τη συνθήκη. Εγώ θα έλεγα ότι κρύφτηκε πίσω από την παλιά συνθήκη. Γιατί με τη νέα πλέον συνθήκη της Λισαβόνας τα κράτη-μέλη έχουν περισσότερες ευθύνες. Όντως, λοιπόν, με τις εθνικές δηλώσεις, αλλά και τις εκθέσεις πεπραγμένων, οι δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νομίζω ότι υπάρχει εδώ ίδια ανάγκη οι επίτροποι να αναλάβουν την πολιτική τους ευθύνη, όπως επίσης και τα κράτη-μέλη. Νομίζω θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ριζοσπάστες εδώ και όχι να δεχθούμε τα μικρά βήματα βελτίωσης. Αυτά ήταν τα λόγια ενός νεαρού Ολλανδού λέοντος, λέει ο πρόεδρος. Τώρα δεν ξέρω να απαντήσει πρώτα ο Επίτροπος γιατί του έγιναν και άλλες ερωτήσεις και μετά να κλείσει ο συγητής μας. Πώς το βλέπετε. Κύριε Επίτροπε, παρακαλώ. Uh, actually, uh, the most of uh, interventions were more comments Ναι, τα περισσότερα σχόλια για το θέμα είναι καλά και νομίζω ότι ο κύριος Φλέινερ ανέφερε το θέμα, ένα θέμα ουσίας. Αυτό το σύστημα των υπογραφών πρόκειται για μια προσέγγιση που θα θέλαμε να ακολουθήσουμε εμείς στην Επίτροπη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ως πρώτο βήμα να έχουμε τις ετήσιες εκθέσεις διαχείρισης με όλα τα θέματα που προσδιορίζονται ε, στο κείμενο που σας παρουσιάστηκε. Ναι, μ' αρέσει η δήλωση των κάτω χωρών, αλλά ακόμα και η δήλωση των κάτω χωρών δεν αντικατοπτρίζει πλήρως αυτό που απαιτείται ε, για την δήλωση αξιοπιστίας, για την Επιτροπή. Πρέπει λοιπόν να εργαστούμε πάνω στο θέμα αυτό και καμιά φορά δεν είναι τόσο ευχάριστο και, ε, και ε, πολιτικά πρέπει να ζητούμε την υπογραφή του Υπουργού αν υποθέσουμε ότι ε, υπογράφει ο, ο, ο, ο υπουργό, αλλά ότι δεν έχει γίνει η βασική εργασία για, το, για την αξιοπιστία, για να υπάρξει η δήλωση αξιοπιστίας. Είναι καμιά φορά δύσκολο για τον υπουργό. Νομίζω ότι αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό είναι τα ουσιαστικά στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται στην έκθεσή μας να καλύπτονται και όλα αυτά τα ουσιαστικά στοιχεία να αντικατοπτρίζονται στο σχέδιο δημοσιονομικού κανονισμού και εδώ θα ήθελα να ζητήσω την πλήρη υποστήριξή σας για να πείσετε το Συμβούλιο να υιοθετήσει το άρθρο 56 του σχεδίου δημοσιονομικού κανονισμού έχει, διότι θα πρέπει να ξέρουμε ότι ε, κάτι θα γίνει στο Συμβούλιο, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί συζήτηση ακόμα στο Συμβούλιο σε σχέση με το άρθρο αυτό. Όταν προσδιοριστεί το θέμα αυτό της ουσίας και της ποιότητας των δηλώσεων αυτών καθεαυτών, θα μπορούμε να συζητήσουμε το επόμενο βήμα το, α, της πολιτικής, κάποιας πολιτικής έγκρισης. Κατά τη γνώμη μου αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να προχωρήσουμε. Σε σχέση με την έκθεση ετησίων, την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων. Και εδώ Νομίζω ότι η δημοκρατία είναι καλό πράγμα, είναι δυνατόν να έχει κανείς διαφορετική, αποκλίνουσα γνώμη. Και η θέση της Επιτροπής είναι ότι οι αιτήσει εκθέσεις δραστηριοτήτων αν έχουν υπογραφεί σε υψηλό διοικητικό επίπεδο επιβάλλουν κάποια ευθύνη πάνω στους διευθυντές να συμπεριφέρονται με ποιοτικό τρόπο. Και αυτό ξέρετε ότι εισήχθη αρκετά πρόσφατα με την μεταρρύθμιση Κίνοκ και αυτό ήταν ίσως από τα βασικά σημεία. Πώς οι διευθυντές να γίνουν πραγματικά υπόλογοι υπεύθυνοι, διότι πριν από την μεταρρύθμιση το θέμα ήταν ότι παρόλο που υπήρχε κάποια πολιτική ευθύνη, στην πραγματικότητα κανείς δεν ήταν υπεύθυνος και υπόλογος. Αυτό είναι το πραγματικό θέμα και αυτό είναι το οποίο προσπαθούμε να προωθήσουμε και είναι σημαντικό. Γενικό Γενικός Διευθυντής να ενημερώνει πλήρως τον Επίτροπό του για το περιεχόμενο της έκθεσης της δραστηριοτήτων και για τις επιφυλάξεις τις οποίες είχε και όλα αυτά να περιληφθούν στις τροποποιημένες οδηγίες προς το Γενικό Διευθυντή και θα θέλαμε επίσης να έχουμε πιο ενδελεχείς ε, πληροφορίες για τις αναστολές και διακοπές. Αυτό είναι σημαντικό μέρος και επίσης οι ανακτήσεις που έχουν γίνει από το Γενικό Διευθυντή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βελτιώσουμε, να βελτιώσουμε πράγματι την ποιότητα των ετησίων αυτών εκθέσεων και νομίζω ότι με τις τροπολογίες αυτές νομίζω ότι θα έχουμε εκθέσεις πολύ καλύτερης ποιότητας. Αυτά ήταν, ε, αυτές είναι ερωτήσεις που μου τέθηκαν και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαίρετη, την αγαστή συνεργασία την οποία είχαμε και τις πολύ καλές προτάσεις και ιδέες για την βελτίωση της διαχείρισης του ευρωπαϊκού χρήματος, διότι είναι και τα, αυτά τα χρήματα των φορολογουμένων μας και θα πρέπει να την χάνουν καλής διαχείρισης. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Έχουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Θέλει το λόγο και η κυρία Μακοβάη και ο κύριος Φέλνερ. Πολύ σύντομα θα σας αφήσω, αλλά μετά ο συγητής. Κυρία Μακοβέη. Thank you, Chair. Um, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, προετοιμάζω τροπολογίες και έχω μερικές συγκεκριμένες ερωτήσεις στον εισηγητή σε σχέδιο με το σχέδιο έκθεση σε σχέση. πρώτον για την παράγραφο 9 Υπάρχουν ειδικέ περιπτώσεις ε, για ε, την μείωση του ποσοστού σφαλμάτων. Η δεύτερη ερώτηση σε ειδικέ συγκυρίες. Ε, πώς θα γίνει η επιστροφή χρημάτων στα κράτη-μέλη ενώ εκκρεμούν στην, παρά, στην παράγραφο 19 ενώ εκκρεμούν οι διορθώσεις, δημοσιονομικές διορθώσεις σε σχέση με την παράγραφο 38 ε, ζητά εξωτερική ανασκόπηση όλων των IAC και γιατί αυτό να μην γίνει από το ελεγκτικό συνέδριο είναι η ερώτηση. Η τέταρτη ερώτηση σχετίζεται με την παράγραφο 79 εάν ε, δεν ε, ακολουθηθεί η απαλλαγή ε, πώς αυτό έχει σχέση με την απαλλαγή και με ποιο θέμα ακριβώς αυτό το οποίο προτείνεται εδώ. Και η τελευταία ερώτηση ε, σε σχέση με την παράγραφο 129, ο ρόλος του αξιολογητή επίδοσης. Αντί να δημιουργούμε μια νέα θέση και πρόσθετη έκθεση, μήπως αυτή η άσκηση δεν θα έπρεπε να ενσωματωθεί στην εργασία της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ευχαριστώ κύριε Φιέλνερ. Ευχαριστώ πολύ. Ακούγοντας τον Επίτροπο ε, θυμήθηκα ότι ξέχασα κάτι εγκάρσιο για όλο το σημείο Δέλτα, για όλο το κεφάλαιο. Και μια ε, που είχα επικρίνει τον κύριο Χατζημαρκάκη, θέλω να το βγάλω αυτό από πάνω Ε, έχει τάση ο εισηγητής να παραπέμπει τα θέματα αυτά στο δημοσιονομικό κανονισμό και θέλει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αλλάξει τους αντίστοιχου δημοσιονομικούς κανονισμούς. Εμείς ε, έχουμε την αίσθηση ότι το αντιμετωπίζουμε λάθος τρόπο. Έχουμε πρόταση για το δημοσιονομικό κανονισμό και έχουμε και ευθύνη για το πώς θα το προωθήσουμε. Ε, ο στόχος μας δεν είναι στην έκθεση της απαλλαγής να αναδιατυπώσουμε το δημοσιονομικό κανονισμό. Αλλού θα το κάνουμε στο οικείο πλαίσιο όχι μέσω της απαλλαγής. Ας πούμε το σύστημα διακοπής και στη συνέχεια αναστολής πληρωμών χωρίς εθνικές ε, δηλώσεις διαχείρισης. Αλλά, ε, συμφωνώ επί της ουσίας, αλλά δεν θα πρέπει να είναι αυτό όρος και προϋπόθεση για να δώσουμε ή όχι την απαλλαγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θεωρώ ότι είναι η σωστή προσέγγιση αυτή. Ας μην αναμειγνύουμε λοιπόν τη διαδικασία αυτή της απαλλαγής με το δημοσιονομικό κανονισμό. Άλλο πράγμα είναι. Ευχαριστώ. Γιώργο, άκουσες τον Επίτροπο να απαντά, άκουσες τους συναδέλφους να ρωτούν, μπορείς να ολοκληρώσεις τώρα εσύ. Θα ήθελα να απαντήσω στη Στάφη Μακοβάη. Όχι όλες, θα απαντήσω στην πρώτη ερώτηση ίσως ρωτήσετε για τις ειδικές συνθήκες της παραγράφου 9. Είσαι η κυρία Κάγιου Λάιτε θα είναι σε θέση να μας πει γι' αυτό. Το 2009 δεν είναι τόσο πολύ δαπάνε στις κύριες χώρες δαπάνης συνοχής που ήταν αντικείμενο ερευνών. Δείγμα, δείγματα είχαμε. δείγματα αφορούσαν κυρίως τις μικρές χώρες που ήταν ε, συγκεντρωτικές. Ισπανία, Γερμανία και οι άλλες ομοσπονδιακές χώρες είναι πιο δύσκολο να γίνει αυτός ο έλεγχος. Δεν ξέρω αν έχω δικαίωμα να το πω αυτό, αλλά νομίζω ε, δείγματα ήταν Δανία, Ισθονία, Ουγγαρία νομίζω, ναι. Οι, αυτοί που δαπανούν τα πολλά όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, για αυτές δεν έγινε ειδική έρευνα. Γι' αυτό έχουμε ειδικέ συνθήκες και γι' αυτό το ποσοστό ασφάλματος μειώθηκε. Πάντως έχουμε και κάτι θετικό. Το θετικό είναι ότι οι διακοπές στην ροή των κεφαλαίων ήδη έγιναν. Δηλαδή έγινε η διακοπή της ροής και γι' αυτό ε, ρώτησα εκ μέρου σα ως τον Επίτροπο να μας δώσει ένα κατάλογο αυτών των διακοπών που χρησιμοποίησε η Επιτροπή ως εργαλείο όχι για να τιμωρήσει αλλά για να πει στις χώρες μέλη διορθώστε την κατάσταση αυτή. Γι' αυτό έχει νόημα να έχουμε έναν ειδικό κατάλογο και ειδικέ συνθήκες. Παράγραφο 19. Τι διορθώσεις μπορούν να γίνουν. Γι' αυτό ζητάμε την πώς λειτουργεί το σύστημα ανάκτησης των κονδυλίων αναφέρθηκα έμεσα στις παρατηρήσεις μου. Κατά κάποιο τρόπο πείτεται διπλά ο Πρώτα, η Επιτροπή, το Λυτικό Συνέδριο και τα κράτη-μέλη εντοπίζουν ένα σφάλμα, τη μη επιλεξιμότητα ας πούμε. εδώ κάτι δεν πάει καλά με το πρόγραμμα αυτό. Και μετά η Επιτροπή θα πει, ναι, ανακτήστε το με ένα άλλο πρόγραμμα. Στην πραγματικότητα Ε, η ανάκτηση αναφέρεται σε ένα μικρό ποσό, αλλά οι διορθώσεις έχουν γίνει. Και γι' αυτό πρέπει να συζητήσουμε το πώς θα ελέγχουμε καλύτερα το θέμα του συνολικού ποσού και δεν είναι εύκολο η Επιτροπή να μας δώσει απάντηση. Ένα λάθος πρόγραμμα ανακτάται με ένα άλλο λάθος πρόγραμμα και δεν πληρώνει ο δικαιούχος, στην περίπτωση αυτή πληρώνει η κυβέρνηση. Δεύτερη φορά λοιπόν πληρώνει ο φορολογούμενος. Πρέπει να προσέξουμε λοιπόν αυτές τις εκκρεμεί διορθώσεις, όπως τις λέμε. Παράγραφος 37. Μια παλιά συζήτηση αυτή. Αν είχαμε μία μεθοδολογία, όλα τα πράγματα θα ήταν εύκολα. Δεν χρειάζεται να ξανά σας αναφέρω τα τη συζήτησης αυτής. Η Κομισιόν δεν κάνει τη μέθοδο της ε, άμεσης φωτογράφησης όπως λέμε που κάνουν οι ελεγκτές. Οι ελεγκτές εφαρμόζουν τη μέθοδο αυτή, τη φωτογραφική α την πούμε μέθοδο για μία χρονιά μόνο. Διαφορετική μεθοδολογία. Αυτό τον εσωτερικό έλεγχο που εφαρμόζει η Κομισιόν δεν μπορεί να την κάνει το ελεγκτικό συνέδριο. Είναι δύο διαφορετικέ μέθοδοι. Επόμενη ερώτηση, η η απόδοση των ελέγχων. Στην πρώτη συζήτηση που είχαμε με τον Επίτροπο Σεμέτα αναφέρθηκε η πρόταση ο εσωτερικός ελεγχτής να επιφορτιστεί με το έργο αυτό. Για μας, ως Ευρωκοινοβούλιο, είστε ελεύθεροι, δεν θέλουμε να παρεύουμε στα εσωτερικά σας. Το θέμα δεν είναι να δημιουργηθεί μια νέα θέση υπαλλήλου, είναι να δημιουργηθεί μια νέα θέση ευθύνης την ευθύνη η συνθήκη την δίνει στην Κομισιόν. Και το θέμα είναι πώς η Κομισιόν θα φέρει σε πέρας αυτή την ευθύνη. Για μένα το πιο σημαντικό είναι το ελεγκτικό συνέδριο ενδέχεται να έχει ένα νέο ρόλο. Διότι ο έλεγχος απόδοσης είναι χρήσιμο ένα πρόγραμμα, είναι αποδοτικό ένα πρόγραμμα, είναι αποτελεσματικό στην εφαρμογή του, είναι έντονα πολιτικό. Το ελεγκτικό συνέδριο λοιπόν αν αξιολογήσουν αυτή την έκθεση αξιολόγησης μπορεί να γίνει ένα λίγο περισσότερο πολιτικό σώμα και μπορεί να αλλάξει η συζήτηση που γίνεται εδώ. Γιατί επαναλαμβάνω το θέμα αυτό έχει έναν έντονο πολιτικό χαρακτήρα. Χρειά. Πολύ περισσότερο πολιτικό από τεχνικό. Οπότε το ελεγκτικό συνέδριο γι' αυτό η αλλαγή είναι πολύ πιο μεγάλη από ό,τι για την Κομισιόν. Δεν είναι λοιπόν, δεν συζητάμε για μια νέα θέση υπαλλήλου, συζητάμε για μια νέα θέση ευθύνης. Ένα σχόλιο σε αυτό που είπε η κυρία Ιβάνοβα για τα ε, αποτελεσματικά συστήματα ελέγχου. Τα κριτήρια για έναν καλύτερο έλεγχο στηρίζεται με βάση τρεις συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου ζητήσαμε πρώτον τις νέες, όχι νέες τις πάντων, την διαχειριστικές δηλώσεις των κρατών μερών όπου εκεί υπάρχουν πολλά κριτήρια που, πρέπει, που, θα, θα βελτιώνανε το σύστημα ελέγχου. Ένα είναι αυτό από τα τρία. Το δεύτερο είναι κατευθυντήρες γραμμές για την απλοποίηση και το τρίτο είναι τα κριτήρια για την διακοπή παροχής. Αν τα συστήματα ελέγχουν δεν λειτουργούν, χρειάζεται διακοπή. Και συμφωνώ με αυτό που είπε η συνάδελφος για την απάτη. Το θέμα απάτη καλύπτεται από αυτά που είπε ο Επίτροπος Σεμέτα όταν είπε υπάρχουν ε, περιοχές, ας το πούμε, και χώρες υψηλού κινδύνου που μπορεί να αναμένουμε περισσότερες απάτες από ό,τι αλλού. Ίσως τα συστήματα ελέγχου των υπηρεσιών της Κομισιόν θα μπορούσαν να βελτιωθούν ή να προσαρμοστούν αντίστοιχα. Κρίστοφερ αναφέρθηκε στο θέμα προσωπικό, προσωπικού υπάλληλοι. Φυσικά το λάβαμε υπόψη μας στην έκθεση. Είναι αυτό που ανάφερε η κυρία Γκρέσλε. Πρέπει όμως να δούμε και την αναλογικότητα. Γιατί είναι λιγότερο από το 5% του προπολογισμού που πάει για το προσωπικό. Πολύ περισσότερο είναι για τη γεωργία, τη συνοχή και πρέπει να το δούμε αναλογικά το θέμα. Και θα πρέπει να δίνουμε τη σωστή μάχη στη σωστή στιγμή και στον κατάλληλο τόπο και αυτό το ανάφερε και η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Να το λάβουμε υπόψη μας, αλλά δεν είναι ένα μείζον σημείο. Ευχαριστώ ιδιαίτερα και τον Επίτροπο Σεμέτα και τους συναδέλφους σας, τον κύριο Χάμ και τον κύριο Άντορν, γιατί είχαμε πολύ καλές συζητήσεις μεταξύ μας. Κρίστοφερ και Γιάν, όπως μας ακούσει κανείς, φαίνεται ότι συμφωνούμε, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα. Θυμάμαι μια συζήτηση που είχαμε που η σύμβολή μου μου έδωσαν ένα χαρτί και μου είπανε μην είσαι τόσο εκνευρισμένος, πιο ήρεμος, πιο ήρεμος. Είχαμε λοιπόν σκληρές συγκρουσιακές συζητήσεις και σας συγχαίρω για το νέο πνεύμα. Βλέπω ότι έχουμε μπροστά μας θετικά βήματα να έχουν γίνει. Και ξαναγυρίζω στο θέμα της ευθύνης και της αξιοπιστίας. Η αξιοπιστία της Ένωσης έχει πέσει πάρα πολύ δυστυχώς και δυχώς οι μέθοδοι δαπάνης στα κράτη-μέλη ουσιαστικά στρέφονται ως κατηγορία κατά της Ένωσης. Όμως αυτοί εκτελούν την δαπάνη των κονδυλίων και γι' αυτό η συζήτηση πρέπει να έρθει στο επίπεδο των κρατών μελών και ο μόνος τρόπος να φέρουμε τη συζήτηση στα κράτη-μέλη είναι δακτυλοδεικτώντας τους ενόχους. Δυστυχώς είναι η μόνη μέθος. Αν ο Βρετανικός τύπος, Φερρυπίν, δει ότι όλα τα προγράμματα του 2010 διεκόπησαν, θα προσπαθήσουν να το δημιουργήσουν βρετανικό θέμα, να γίνει ένα θέμα συζήτηση στη Βρετανία. Και έγινε αυτό με του Financial Times και χαίρομαι γι' αυτό, αλλά για να το κάνουμε αυτό, να μεταφέρουμε τη συζήτηση στο εθνικό πλαίσιο, χρειαζόμαστε διαφάνεια, πίνακε, νούμερα. Γι' αυτό όλα αυτά τα έξι αιτήματά μας είναι στο στάδιο ότι εμπεριέχουν αυτό το αίτημα για περισσότερη διαφάνεια. Η Κομισιόν από πέρυσι ξεκίνησε με το βιβλίο εδώ, το, σας το δείχνω, όπου αναφέρει ονομαστικά συγκεκριμένε χώρες και αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Ευχαριστώ και το Ελληνικό Συνέδριο γιατί είχαμε πολύ σοβαρές και σε βάθος συζητήσεις μαζί τους. Σας συγχαίρω για το νέο ρόλο σας που όπως είπα θα είναι πιο πολιτικός από εδώ και μπρος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σίγητα. Και ο κύριος Φιένερ σας χειροκρότησε ή δεν ξέρω σας επιφήμισε. Ε, μόλις μπήκε η κυρία Τσέσκοβα και θέλει κάτι να πει. Παρακαλώ. Ε, ε, ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Τα όσα άκουσα, ε, όλα αυτά τα προσυπογράφω, τα υποστηρίζω. Μιλήσατε για τα κράτη-μέλη και αυτό είναι κρίσιμο. Αλλά έχω μια μικρή παρατήρηση. Ελπίζω ότι θα με καταλάβετε. Όταν μιλήσατε, μιλήσατε για την υπευθυνότητα των κρατών μελών. Μιλήσατε για τις εθνικές στατιστικές και μιλήσατε για το ε, πώς ε, κάνουν τις αναφορές τους στα κράτη-μέλη και μετά είπατε και κάτι άλλο. Είπατε ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα κράτη όπου ξέρουμε ότι μπορεί να υπάρχουν σφάλματα, ε, σφάλματα ή λάθη αναμένονται. Ε, δεν συμφωνώ πλήρως με αυτό, διότι πιστεύω ότι στο Κοινοβούλιο και σε αυτή την Επιτροπή κάθε χρόνο βλέπουμε ότι το ποσοστό λαθών, σφαλμάτων, και, και αυτό το οποίο οφείλεται στην απάτη μπορεί να διαπιστωθεί σε διαφορετικά κράτη-μέλη, σε όλα τα κράτη-μέλη. Ίσως με διαφορετικό τρόπο θα ήθελα συνεπώς να επισημάνω ότι κάτι το οποίο δεν συζητούμε σήμερα, όταν μιλάμε για την απαλλαγή για το 2009 είναι κάτι που δεν θα μπορούσαμε ίσως να συζητήσουμε του χρόνου, διότι ίσως να ήταν σημαντικό του χρόνου. Πιστεύω ότι εμείς ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προβλέψουμε όταν ε, ανοιχνεύουμε σφάλματα και λάθη και όταν εξετάζουμε την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε ότι μερικά κράτη-μέλη θα έχουν προβλήματα στο μέλλον και πρέπει αυτό να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την έκθεση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο επίσης. Και θα ήθελα να πω ότι ε, συμφωνώ, αλλά ε, ένα συνάδελφος είπε ότι πρέπει να ευχαριστούμε πάντοτε τον εισηγητή, αλλά εγώ το εννοώ όταν τον συγχαίρω και τον ευχαριστώ. Μπράβο σας. Λοιπόν, ολοκληρώνεται έτσι το σημείο 7 και για λόγους τάξεως πρέπει να σας πω ότι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών λύγει τη Δευτέρα 7 Μαρτίου, σε μια εβδομάδα δηλαδή ακριβώς, στις 12 η ώρα το μεσημέρι και θα ψηφίσουμε στις 28 του μηνός Μαρτίου εδώ στις Βρυξέλλες. Παίρνουμε τώρα στο σημείο 8. Θα είναι συντομότερο, πιστεύω. Είναι όλες οι ειδικέ εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Έχουμε πάρα πολλά έγγραφα εργασίας εδώ, τα οποία εγκρίναμε ή τουλάχιστον τα συζητήσαμε. Και παρακαλώ τον εισηγητή κύριο Χατζημαρκάκη να μας πει σύντομα δύο λόγια όμως γι' αυτό ακόμα. Ναι. Στα γερμανικά τώρα νομίζω είναι πάρα πολύ σύντομο. Μπορούμε να διεκπαιρεώσουμε πολύ ε, γρήγορα. Θα βρείτε την έκθεσή μου στο σημείο 8 και θα δείτε από τα περιεχόμενα ότι πρόκειται για 11 ειδικέ εκθέσεις. Ε, υιοθετήσαμε τις συστάσεις των ε, συναδέλφων, οπότε δεν υπάρχει και καμία αλλαγή που έκανα εγώ και είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις. Ο Πρόεδρος. Θέλει να πει κανείς τίποτα για αυτά τα θέματα, όχι. Ωραία. Το ίδιο ισχύει ως προς την προθεσμία κατάθεση τροπολογιών και για την έκθεση αυτή, 7 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι και θα ψηφίσουμε στις 28. Ερχόμαστε τώρα στη δική μου έκθεση. Τώρα είμαι λίγο στριμωγμένος γιατί ε, είμαι και εισηγητής και πρόεδρος και έχουμε άλλους πρόεδρους, μας τελείωσαν. Ποιος είναι εδώ ο πρεσβύτερος, όχι στην ηλικία, στη θητεία, στην επιτροπή. Ξέρω ότι είμαι εγώ, αλλά πρέπει να ε, παρουσιάσω και την έκθεσή μου. Μετά από μένα... κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ για ε, όλο σας το έργο, ε, για τις απαντήσεις σας και θα είμαστε σε επαφή, να μην χαθούμε. Ε, συνεχίζουμε το σημείο 9. Απαλλαγή για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης. Κατέθεσα μια έκθεση την οποία θα μπορούσα να σας παρουσιάσω σε 10 κεφάλαια. Ξέρετε συνάδελφοι ότι είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Ανάπτυξης. Είναι πολλά τα λεφτά. 22,6 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2008 στο 2013. 22,6 δις είναι ε, πολύ περισσότερο από το Ερίνα το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, το φετινό και σας είπα ότι είναι 10 χωριστά τα κεφάλαια ή πώς να το πω αλλιώ, 10 ξεχωριστά στοιχεία τα οποία περιγράφω. Το πρώτο είναι οι παράγραφοι 2, 3 και 4 που κυρίως λένε το εξής. Επαναλαμβάνουμε την κριτική μας για το ότι δεν είναι συμπεριλαμβανόμενο στον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξη. Το ξέρουμε αυτό, δεν έχει συμπεριληφθεί στον προπολογισμό. Αλλά είναι το πιο σημαντικό μέσο για την αναπτυξιακή βοήθεια. Και στις παραγράφους 2, 3 και 4 υποστηρίζω αυτά που είχαν υποθεί προηγουμένως και που είχε δηλώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θέλει να εγγράψει στον προπολογισμό και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη ε, και γίνεται μια έκκληση και μια παρότρινση εδώ και προς τα κράτη-μέλη και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2014 και μετά να ε, έχει ενταχθεί στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη. Στη συνέχεια. Γι' αυτό θα ενδιαφέρει κυρίως την κυρία Χόλμαγερ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί το 20% της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας να δίνεται στη βασική ε, παιδεία, στη δημοτική εκπαίδευση και στη βασική υγεία, στην πρωτοβάθμια. Και το ζητάει αυτό και η παράγραφος 2. Άλλο στοιχείο. Αναγνωρίζουμε ότι το ελεκτικό συνέδριο στην έκθεσή του λέει ότι η διαχείριση του 8ου, 9ου και 10ου ταμείου είναι καλή ε, περιγραφή ε, των πεπραγμένων και επί της ουσίας ε, ανταποκρίνεται η κατάσταση ε, όπως περιγράφεται στην πραγματικότητα. Στις παραγράφους 7, 8, 9, 10 και 11 αναφέρω τις ελλείψεις και τα προβλήματα που τα επισημαίνει και το ελεγκτικό συνέδριο. Και το θέμα είναι ότι η δήλωση αξιοπιστία δεν αφορά τη διευκόλυνση επενδύσεων τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά αυτή έχει μπει σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, αλλά υπάρχει μια αδυναμία στο συνολικό δημοκρατικό έλεγχο. Παράγραφος 12 έως και 17. Αυτό έχει να κάνει με το λογιστικό σύστημα. Ε, έχει διαπιστωθεί κάποια βελτίωση εκ των υστέρων έλεγχη του Europe Aid ε, κάνει δουλειά το EuroPaid και οι διάφορες αντιπροσωπείες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε αυτές τις παραγράφους λοιπόν αναφέρομαι σε αυτό το θέμα. Επόμενο στοιχείο, η παράγραφος 18 είναι η συνέχεια που δίδεται στη συγκεκριμένη ειδική έκθεση ε, για την Ανατολική και Δυτική Αφρική. Ε, επόμενο στοιχείο, κάπως δύσκολο και ακαθόδες τώρα και σωστά το επεσήμενε και η κυρία Γκρέσλε είναι η παράγραφος που αναφέρεται ε, στους τόκους. Τι θα τους κάνουμε τους τόκους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Πραγματική υποστήριξη, ε, μόνο ως δαπάνης υποστήριξης, το λέμε αυτό, στην παράγραφο 19 και δεν είναι θέμα χρηματοδότησης του ε, προσωπικού ή μισθοδοσίας του προσωπικού. Ε, αυτό παραμένει προσυζήτηση όμως και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επόμενο σημείο, ε, τέσσερις παράγραφοι, 20 έως και 23. Είναι η όλη προβληματική της δημοσιονομικής ενίσχυσης του προϋπολογισμού. Στο μεταξύ έχει εκδοθεί μια πράσινη βίβλος όπου πιστεύω νομίζω την επόμενη Πέμπτη θα το συζητήσουμε γιατί πρέπει να γνωμοδοτήσουμε στην ε, Επιτροπή Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Νομίζω ότι όλο το σύστημα της υποστήριξης χρηματοοικονομικής βοήθειας ε, του προϋπολογισμού πρέπει να αλλάξει στον έλεγχό του. Όχι μόνο το input, δηλαδή πόσα λεφτά δίνουμε, αλλά και η ποιότητα και εκ του αποτελέσματο να κρίνεται και να ελέγχεται. Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο ρόλο των αντιπροσωπιών στην ενίσχυση του προσωπικού εκεί και επίσης γίνεται αναφορά σε ένα μέσον που χρησιμοποιεί η Παγκόσμια Τράπεζα για που λέγεται ΠΕΦΑ, που είναι ε, δημόσιες δαπάνες και η, ε, οικονομική λογοδοσία για μεγαλύτερη διαφάνεια. Ε, άλλο στοιχείο που θέλω στην έκθεση είναι οι στρατηγικές ελέγχου της Europaid και πάλι. Πρέπει να εφαρμόζονται ε, και να ελέγχονται καλύτερα, 34 και 35 παράγραφοι είναι αυτοί. Και ένα τελευταίο, παράγραφοι 36 έως και 45 είναι η επενδυτική διευκόλυνση, η Investment Facility της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Τρέχουν διάφορα προγράμματα εκεί, ε, αλλά πιστεύω ότι οι εκπρόσωποι ε, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι παρόντες κιόλας εδώ. Νομίζω ότι μέρα με τη μέρα βελτιώνεται η κατάσταση, αλλά θα πρέπει να έχουμε καλύτερη συνεννόηση και συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θέλω μεγαλύτερο πλαίσιο συνεργασίας και ε, μεγαλύτερη συνεννόηση και ενόψη της απαλλαγής και ζητώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να δείχνει μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς το μαύρο κατάλογο των ε, απαταιώνων. Λίστα απαταιώνων ε, στις παράγραφο 42 το αναφέρω αυτό Ξέρουμε ότι υπάρχει μια υπόθεση ενός πρώην υπαλλήλου της Όλαφ και ζητώ πιο τακτική αναφορά στην Επιτροπή μας. Μια φορά το χρόνο νομίζω δεν φτάνει. Χρειάζεται έτσι λίγο πιο τακτική επαφή και πιο διαρθρωμένη συνεργασία. Αυτά είναι λοιπόν τα 10 σημεία, τα 10 κεφάλαια που σας είπα, ε, στα οποία αναφέρομαι στην έκθεσή μου. Και καλώ τους συναδέλφους να δώσουν τα σχόλιά τους. Δεν ξέρω, θέλει το λόγο και το ελεκτικό συνέδριο. Θέλει κανείς το λόγο από τους εκπροσώπους του ελεκτικού συνέδριου. Όχι. Πείτε μας κάτι κι εσείς. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω άλλη μια φορά ότι ε, η έκθεσή σας αντικατοπτρίζει πάρα πολύ ορθά τις ε, διαπιστώσεις μας ε, και η έκθεση υποστηρίζεται, εγκρίνεται. Ευχαριστώ. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει το λόγο. Θέλει. Η ε, κυρία Τσέσκοβα και ο κύριος Έπινγκ από συναδέλφους. Άλλος κανείς. Α, θέλετε κι εσείς, ε, η κυρία Χολμάγερ. Καλώς. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, και η κυρία Γκρέσλε. η Επιτροπή όμως πρώτα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα ε, πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον πρόεδρο και εισηγητή για την έκθεση. Χαιρετίζουμε αυτήν την έκθεση θα ήθελα να ε, επιβεβαιώσω τα όσα είπε ο Επίτροπος για την ε, απαλλαγή ε, υποστηρίζει, εγκρίνει την έκθεση ένα από τα θέματα που τονίστηκε στην έκθεση απαλλαγής είναι η ανάγκη να υπάρξουν δείκτες για, τον, για το κατάλοιπο κινδύνου σχετικά με τα σφάλματα, τον υπολοιματικό κίνδυνο. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο αναφέρεται στην έκθεση εισήγηση είναι το θέμα του προϋπολογισμού βεβαίως, όπου η Επιτροπή χαιρετίζει τις διαπιστώσεις ε, και θεωρεί ότι όλα βαίνουν προς την σωστή κατεύθυνση ε, και υπάρχει καλύτερη τεκμηρίωση για τις εκταμιεύσεις ε, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Σημείο 33 του σχεδίου ψηφίσματος θέτει το θέμα μιας δήλωσης εξάντε για τις δικαιούχους χώρες. Αναφερθήκατε στην αξιολόγηση ΠΙΒΑ για την συζυγήσεις λογοδοσίας με βάση το 33. Θα το θεωρήσουμε ως βάση για την δήλωση αξιοπιστίας. Είναι βασικό εργαλείο και πιστεύουμε με άλλους ε, δωρητές ότι είναι καλύτερη βάση να έχουμε ανεξάρτητη γνωμοδότηση για την ε, ανεξάρτητη ε, πορεία των, της διαχείρισης. Αυτές οι δηλώσεις δημοσιοποιούνται και μετά συζητούμε για τις συστημικές αδυναμίες που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Θα εξακολουθήσουμε να ασχολούθαμε με το σύστημα σε σχέση με τα συμφέροντα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για την διοικητική υποστήριξη. Εδώ η νομική βάση είναι αρκετά σαφής. Αυτοί, αυτοί οι τόκοι EDF δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το κόστος του μόνιμου προσωπικού. Αλλά είναι σαφές από τη νομική βάση ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι τόκοι EDF του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης ε, για υποστήριξη διοικητική. Νομίζω ότι θα σταματήσω εδώ και θα επανέλθω ίσως αργότερα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ακολουθήσω τη σειρά και το μέγεθος των πολιτικών ομάδων. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, πρώτη σκιοδησηγήτρια, η κυρία Χολμάγερ. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αλλά και εισηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις καλές ε, συζητήσεις που είχαμε. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ για την έκθεση, την καλωσορίζω και στα περισσότερα σημεία τη συμμερίζομαι. Ιδιαίτερα και θέλω να το πω από την αρχή, θεωρώ απολύτως πήγον από το 2014 και μετά η Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Βοήθεια και ό,τι άλλο κάνουμε σε αυτό το τομέα και όλη η χρηματοοικονομική πόροι στο τέλος ε, από το 2014 και μετά να ε, είναι τμήμα του κανονικού κοινοτικού προϋπολογισμού και όχι σε έκτακτη διαδικασία. Είναι πάντα προβληματικό να έχει κανείς έκτακτες περιστάσεις, έκτακτους ε, προϋπολογισμούς που διαφεύγουν της πλήρους εποπτείας και ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό εμποδίζει και τη συνέπεια και τη συνέχεια της πολιτικής και στην πράξη. Θα ήθελα να βρεθώ σε δύο-τρία σημεία που θεωρώ πολύ σημαντικά στην αναπτυξιακή βοήθεια. Πρώτον, ε, θεωρώ ότι στην αναπτυξιακή βοήθεια νομίζω ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη κάλυψη, ένα κατακαιρματισμό, ε, μια πολύ μεγάλη διασπορά και των τομέων που μας ε, απασχολούν αλλά και των χωρών δεν θα είμαστε σε θέση ε, όλες τις χώρες που βασανίζονται και υποφέρουν και ζουν σε να τις υποστηρίζουμε ε, με το σωστό τρόπο ή στο επίπεδο που χρειάζονται. Θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητες και κέντρα βάρους. Και χαίρομαι γιατί το ανέφερε ήδη στην Επιτροπή μας και ο Επίτροπος Πίμπαλξ ότι θα πρέπει στη γεωργία, στην υγεία, στην παιδεία να έχουμε κάποιες προτεραιότητες απέναντι σε διάφορα άλλα προγράμματα που μπορεί να είναι καλοπροαίρετα αλλά τελικά δεν ανταποκρίνονται στους στόχους ε, της ανάπτυξης, ε, της αηφορίας και της ε, αυτάρκειας ενός κράτους. Κάτι που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση τώρα σε σχέση με όλα αυτά. Αν δούμε τι συμβαίνει στη Βόρεια Αφρική αυτό τον καιρό και τις εξελίξεις θα πρέπει να μας απασχολήσει και το θέμα της βοήθειας της Μεσογειακής και πώς θα βοηθήσουμε τις χώρες αυτές να οικοδομήσουν δομές και οικονομικές και δημοκρατικές. Γιατί μέχρι τώρα η ε, ε, κυβερνήσεις ε, ήταν ε, αυταρχικές, οι οποίες τώρα ε, εκλείπουν και αν μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε στη θετική κατεύθυνση θα πρέπει να είναι απόλυτη προτεραιότητα. Γιατί είναι και οι άμεσοι γείτονέ μας οι λαοί αυτοί. Όχι μόνο αυτό, αλλιώς γνωρίζουμε αν αποτύχει τι προβλήματα θα πρέπει να αναμένουμε και στην Ευρώπη, που πλευρά μετανάστευσης. Όταν ο κόσμος δεν έχει στον ήλιο μοίρα, τρέχει στη διπλανή χώρα να βρει την τύχη του. θα, θα πρέπει να τους βοηθήσουμε να παραμείνουν στις χώρες τους για ε, να αναπτυχθούν αυτές μέσω της αναπτυξιακής μας βοήθειας. Είναι πολύ σημαντικός στόχος. Ε, χρειάζεται συντονισμό για να δώσουμε σε μια νέα γενιά μια πιθανότητα μια ελπίδα να βγει από αυτή την απελπισμένη κατάσταση στην οποία ζει σήμερα. Δεύτερο, η δημοσιονομική ενίσχυση. Μακροοικονομική βοήθεια είναι αυτό και πάντα ε, είναι προβληματικό. Εγώ δεν είμαι πάγια αντίθετη με μια δημοσιονομική βοήθεια να δίδεται μόνο εφόσον έχουμε κάποια στοιχειώδη εχέγγυα με προηγούμενη προετοιμασία των προγραμμάτων και εγγύησης από πλευράς των κυβερνήσεων και όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά να είναι υπαρκτές αυτές οι εγγύησει ότι τα χρήματα δεν θα είναι αντικείμενο λαθροχειρίας ή θα πάνε σε λάθος χέρια ή σε λάθος τσέπες σε σχέση με τους πραγματικούς στόχους της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής ε, βοήθειας. Θα πρέπει να υπάρχουν, αν μη τι άλλο, ελάχιστες προδιαγραφές, αλλιώς δεν ξέρω, να βρούμε κάποιον άλλο τρόπο να κάνουμε αναπτυξιακή ε, πολιτική και αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτά. Λίγα είναι αυτά που σας λέω. Τώρα για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τους τόκους. Πού πηγαίνουν αυτοί οι τόκοι, δεν κατάλαβα. Ε, πληρώνουμε μισθού από εκεί, σε πιο προσωπικό. Ε, από πλευράς διαφάνειας, γιατί διάβασα και κάτι ποσά που δεν είναι και ευκαταφρόνητα. Είναι έτσι αρκετά γενναία και σεβαστά. Και είναι ενδιαφέρον να μάθουμε τι γίνονται αυτά. Και πού πηγαίνουν ουσιαστικά και πραγματικά και τι προσφέρουν. Θα ε, με ενδιαφέρει επίσης να δω τι προσωπικό εκεί έχει προσληφθεί, για πόσο διάστημα, είναι με σύμβαση έργου, είναι με σύμβαση αορίστου χρόνου, τι συμβάσεις είναι αυτές. Είναι ένας τρόπος να αντισταθμίζεται η έλλειψη προσωπικού. Πού πηγαίνουν αυτοί οι τόκοι, εν πάση περιπτώσει, χρηματοδοτήσεις μισθών. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή και πάλι και νομίζω ότι θα έχουμε κοινή βάση και μια καλή βάση για την απαλλαγή. Για το 8ο, το 9ο και 10ο παρακαλώ Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Η κυρία Τσέσκοβα. Ε, ε, ναι, παίρνω και πάλι το λόγο, κύριε Πρόεδρε, και θα ήθελα να συνεχίσω τα όσα είπε η προλαλή σα, αλλά θα επικεντρωθώ σε ένα άλλο θέμα. Πρόκειται για το 5 που νομίζω το σημείο 5 που είναι σημαντικό σημείο. 20% των χρημάτων που δίδονται για την ανάπτυξη θα πρέπει ε, να δίδονται, να παρέχονται για την εκπαίδευση και τη δημόσια υγεία. Και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στην, επιτρο... στην γνωμοδότηση της Επιτροπής ΔΕΒΕ, σύμφωνα με την οποία θα έπρεπε να επικεντρωθούμε στην υγεία των μητέρων. Θα ήθελα να, αρχί... να ανοίξουμε μια συζήτηση για το θέμα αυτό εδώ. διότι κυρίως στους τομείς αυτού για τους οποίους παρέχονται τα κονδύλια αυτά για την ανάπτυξη, εκεί οι μητέρες και οι γυναίκες είναι οι ενδιαφερόμενες κυρίως. Ξέρουμε όλοι ότι τα πρότυπα, τα επίπεδα που υπάρχουν εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχουν στις χώρες αυτές. Συνεπώς, Ίσως αυτό το θέμα, το θέμα της υγείας των μητέρων θα μπορούσε να διευρυνθεί, να επεκταθεί για να περιλάβει την, το δικαίωμα στη σεξουαλική, σεξουαλική υγεία και αναπαραγωγική υγεία, διότι ε, υπάρχουν περιοχές όπου θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ε, ε, διευθετήσουμε ή να βοηθήσουμε να διευθετηθούν αυτά τα ειδικά προβλήματα και να παρέχουμε χρήματα και κονδύλια για τα θέματα αυτά. Θα ήθελα ακόμα και υψηλότερο ποσοστό ε, για τα θέματα αυτά, διότι πιστεύω ότι αυτό θα βοηθήσει και αντιστοιχεί στις αξίες που θέλουμε να προωθήσουμε, τις αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού που θέλουμε να προωθήσουμε στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Και αυτό κάνουμε χρηματοδοτώντας με διάφορα κονδύλια, με διάφορα ταμεία, με βοήθεια, με ενισχύσεις που παρέχουμε εκεί. Νομίζω λοιπόν εν ώψη της σύνθεσης του πληθυσμού εκεί και σέβομαι βεβαίως την κουλτούρα τους, αλλά ότι θα έπρεπε να, να λάβουμε υπόψη την κουλτούρα που υπάρχει στην κάθε χώρα και να πούμε ανοιχτά ότι και αυτό είναι το σημείο 6 της γνωμοδότησης. Αν θέλετε να του ρίξετε μια ματιά, η γνωμοδότηση στην οποία αναφέρθηκα της Επιτροπής ΔΕΒΕ, θα μπορούσαμε ίσως να περιλάβουμε εκεί ε, και το δικαίωμα στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. Βεβαίως χαιρετίζω πλήρως και συμφωνώ ότι ίσως όχι 20% αλλά ακόμα και ένα υψηλότερο ποσοστό αυτών των κονδυλίων θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την υγειονομική περίθαλψη και υγεία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω ε, να εξευμενήσω τις ε, γυναίκες συναδέλφους, θα τους δώσω πρώτα το λόγο, οπότε τώρα η κυρία Γκρέσλε. Θέλω να επανέλθω σε αυτό το θέμα των τόκων και των μισθών από τους τόκους. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε ότι θα ήταν, ήταν λέει, τελείως φυσιολογικό κάτι τέτοιο. Έχω αρχίσει και ανησυχώ από την απάντηση αυτή. Από τόκους να πληρώνουμε μισθούς, ναι. Πώς έτσι το Συμβούλιο έχει αντιδράσει με τον ΑΒ τρόπο, γιατί θα πρέπει να ενδιαφέρεται το Συμβούλιο, γιατί είναι αρμόδιο για την εγγραφή αυτού του κονδυλίων στον προϋπολογισμό. Και πώς το γράψαν. Και τώρα τι διδάγματα έχουμε εξαγάγει. Θα είναι στάνταρ ερώτημα στο ερωτηματολόγιο μα ή θα έχει και τίποτα συνέπειε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Ο κύριος Έπινγκ. Eh. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο και εμένα. Με προσοχή διάβασα την έκθεσή σας. Νομίζω ότι ε, διέπεται από μία αδιανοητική ε, τιμιότητα και είναι και νυφάλια έκθεση και αντικειμενική και συγχαρητήρια. Ωστόσο θα ήθελα να σας υποβάλω και κάποιες ε, προτάσεις μου δημιουργικά να συμβάλλω και εγώ στην συγγραφή της έκθεσής σας. Λέει η έκθεση και ισχύει βέβαια ότι το 10ο Ταμείο Ανάπτυξης έχει γνωρίσει αύξηση 64% ε, έχει φτάσει στα 22,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το ένατο. Και η πρώτη ερώτηση που μου έρχεται στο μυαλό είναι υπάρχει αποφυτικότητα αν αυξηθεί τόσο πολύ μια χρηματοδότηση. Κοιτάω τον προπολογισμό για την αναπτυξιακή βοήθεια σε διάφορα κράτη-μέλη και στις περισσότερες περιπτώσεις και πάρα πολύ γρήγορα εξαντλείται η δυνατότητα απορρόφησης. Λεφτά υπάρχουν, θέλουν να τα δαπανίσουν, αλλά δεν μπορούν τα κράτη να τα απορροφήσουν. Και υπάρχει μια πίεση για την απορρόφηση, γιατί όσο προχωράει και ο χρόνος ε, και τελειώνει το έτος, αυξάνεται και η πίεση για να απορροφήσουν άρον-άρον τα κονδύλια. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το πρόβλημα της απορροφητικότητα και θα ήθελα να το βάλουμε και στην έκθεση για να τονίσουμε. Ένα δεύτερο, Βεβαίω δεν θα πρέπει να τρέχουμε ε, και να αποφεύγουμε την επικαιρότητα. Ε, μία από τις προαλήσεις σε συναδέλφους μίλησε για τις εξελίξεις στη Βόρεια Αφρική. Στις 2 Φεβρουαρίου, ενεστώτος έτους, και η κυρία Άστον εδώ, στη Μίνη, ε, Σύνοδο και είπε ότι η πολιτική γειτονία και συγκεκριμένα στη Μεσόγειο είχε αποτύχει. Εντάξει. Σημαντικό αυτό είναι το συμπέρασμα, γιατί τότε μόλις άρχιζαν οι διαδηλώσεις στην Αίγυπτο και οι οποίες οδήγησαν στην αποχώρηση του Μουμπάρακ και ακολούθησαν ε, τα πράγματα και εξελίξεις που γνωρίζουμε. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης είχε εκεί καμία επιρροή στη Βόρεια Αφρική θετική ή καμία ή αρνητική. Ήταν μικρή η συμμετοχή του ανεπαρκής. Δεν θα πρέπει να αποφεύγουμε και την πραγματικότητα να την αντικρίσουμε κατάματα. Γιατί είναι και ε, ένα εργαλείο με ένα μέσο, αλλά θα πρέπει να βλέπουμε πώς λειτουργεί στην πράξη. Κάτι άλλο που θέλω να σας πω, ε, ε, τι, να ρωτήσω μάλλον, τι φρονείτε για τις μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις, NGOs είναι και θέμα εμπιστοσύνη και σχέσεων, γιατί δεν είναι όλες άγιες η ΜΚΟ. Κάπου λέτε ότι είναι πολύ σημαντικές για την αηφόρο ανάπτυξη. Sustainable Development. Στο 6. Μα το 2009 η έκθεση λέει ότι ακριβώς οι ΜΚΟ αυτές έχουν κάποια έργα που δεν είναι αηφόρα. Και πρόκειται για ένα δισεκατομμύριο ευρώ εκεί. Είναι μεγάλα ποσά αυτά. Και η ειδική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου θα πρέπει να ε, αξίζει μεγαλύτερη προσοχή και σημασία. Μια άλλη ειδική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου λέει ότι η ολοκλήρωση στην Ανατολική και στη Δυτική Αφρική ε, δεν ήταν τελείως αποτελεσματική. Ε, για να είμαστε ειλικρινεί, θα πρέπει να πούμε ότι απέτυχε όταν λέει ότι, δεν ήταν, ότι ήταν μόνο εν μέρη αποτελεσματική, άρα μηδέν. Είστε πολύ επικριτικός σε σχέση με πετρελαϊκές εταιρείες ή πολυεθνικές. Δεν είστε το ίδιο επικριτικός με τις ΜΚΟ. Θα πρέπει να κρατήσετε και εσείς αποστάσεις. Αυτό το ονομάζουν κουέγκος οι Αγγλοσάξονες. Ε, και σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική στήριξη, τη μακροοικονομική βοήθεια, άκουσα κριτική προηγουμένως και τη συμμερίζομαι. Σε κάποιες περιπτώσεις δίνουμε χρήματα σε κάποιες χώρες ως μακροοικονομική βοήθεια ε, για να μπορέσουν να τα απορροφήσουν γιατί δεν μπορούν να απορροφήσουν ε, τη διαφορετική μορφή βοήθειας, στην αναπτυξιακή. Ε, θα πρέπει να υπάρχουν πολλά κριτήρια για την ενίσχυση του προπολογισμού. Ξέρω πολλές χώρες στην Αφρική που την χάνουν υποστήριξη χωρίς να έχουν τη διοικητική δομή. Σε ό,τι αφορά τις δικές μας αντιπροσωπείες εκεί, πρέπει να σας πω με κάθε ειλικρίνεια ότι και αυτές είναι εν μέρη αποτελεσματικές. Δηλαδή καθόλου, όπως σας είπα προηγουμένως, αυτό το εν μέρη. Χρειάζεται περισσότερο προσωπικό. Δεν κατάλαβα, η απάντηση σε όλα τα προβλήματα είναι περισσότερο προσωπικό. Ο κύριος Σμιτ, εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής που κατά τα άλλα ήταν συνάδελφός μου στο ιδιαίτερο γραφείο του Επιτρόπου κυρίου Κάλλας και γνωριζόμαστε πολύ καλά και ο ίδιος γνωρίζει τις αντιπροσωπίες, θα μπορούσε να μας ενημερώσει περισσότερο. Δεν ξέρω όμως αν είναι η λύση να αυξάνεται συνεχώς το μέγεθος των αντιπροσωπιών μας για το micromanagement, αυτή τη μικροδιαχείριση. Αυτά ήθελα να σας πω ως συμπλήρωμα μόνο της έκθεσής σας σας τα καταθέτω, εσείς θα κάνετε ό,τι θέλετε. Ε, πάντως μερικά θέματα νομίζω είναι κρίσιμα και χρήσιμα και σε σχέση με την ε, επικαιρότητα. Για να δούμε και τι συμβαίνει στους δρόμους και όχι μόνο στους δρόμους των αραβικών κρατών. Να μην χάνουμε και αυτή την πτυχή της πραγματικότητας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χατζημαρκάκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για την έκθεση. Πολύ καλή βάση για τη συζήτησή μας. Ε, θέλω να μπω σε αυτό το θέμα ακριβώ για τη Βόρεια Αφρική. Δεν είναι μόνο αραβικέ χώρε, είναι η Βόρεια Αφρική ολόκληρη. Το είπε και η συνάδελφο Χολμάγερ. Διερωτάται κανεί πώ μα ξέφυγε έτσι η κατάσταση και η συζήτηση. Είναι λίγο λυπηρό αυτό και θλιβερό. Θα μπορούσαμε κανονικά να είμαστε σε θέση να δώσουμε άμεση βοήθεια τη γειτονία η κυρία Άστον, που τη λένε πλέον κυρία Άψεντ, η κυρία Πούσα, ήταν εξαφανισμένη. Έχουμε κάποιους πόρους στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Πώς μπορούν αυτοί να αναδιαταχθούν, να πάνε σε άλλους σκοπούς. Στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπάρχει αυτή η ευελιξία. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ξέρω αν υπάρχει. Και παρακαλώ να μου απαντήσετε πόσο γρήγορα μπορεί κανεί να διαθέτει πόρου επιγοντε. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τώρα γεννάται το μεγάλο πρόβλημα ότι η Τράπεζα του Αταλή, θυμάστε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότηση και ανάπτυξη, από ό,τι φαίνεται θέλει να ανακατευτεί και στη Βόρεια Αφρική. Βρήκε την ευκαιρία να επέμβει. Και τι στρατηγική έχουν. Γιατί βλέπει ότι είναι καμπή, ότι αλλάζουν τα πράγματα, θέλει να χωθεί και αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καμιά ιδέα. Στην παράγραφο 9 τώρα, βλέπω ότι αναφέρεται την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και αυτούς τους πόρους που εμεί δεν έχουμε λόγο και δεν έχουμε και εικόνα το επικρίνει αυτό ο εισηγητής. Στα γερμανικά η κριτική είναι πάρα πολύ δυσνόητη έτσι όπως έχει μεταφραστεί. Εγώ θέλω να το τονίσω. Δεν το θεωρώ σωστό να μην έχουμε πρόσβαση στο τι κάνει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πολλό δε μάλλον που είναι πολύ διαφανής. Δεν υπάρχει λόγος να μας τα κρύβουν, να μας έχουν απ' έξω από αυτή την ιστορία. Και ένα τελευταίο Δυστυχώ, μόλις βγήκε ο κύριος Χέιστε Φρίς, αλλά ε, υπάρχουν κάποιες εσωτερικές σκέψεις στο Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο για το εξής πρόβλημα και φαινόμενο στη βοήθεια στις θεομηνίες. Πολλά χρήματα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης πηγαίνουν στην ανθρωπιστική βοήθεια για τις θεομηνίες. Και στην αιτία, ας πούμε, σε άλλες χώρες, οι δωρητές κάθονται μεταξύ τους, δίνουν τα λεφτά, αλλά δικαιούχοι δεν έχουν τη δυνατότητα να αποδείξουν ότι πηγαίνουν σε σωστό σκοπό τα χρήματα. Δηλαδή τους επιβαρύνουμε πολύ τους δικαιούχους με τους δικούς μας εσωτερικούς κανόνες. Το σκέφτεται αυτό, λέει το ελεκτικό συνέδριο. Δεν θα μπορούσαμε να δούμε διεθνώς πώς θα το απλουστεύσουμε. Εμείς οι Ευρωπαίοι, μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση για την επίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια σε ομιλίες. Αυτό είναι θέμα της Επιτρόπου κυρίας Γεωργίευα, της Βουλγάρας Επιτρόπου. δεν ξέρω, με μακροοικονομική βοήθεια χωρίς ε, κάποιο λογιστικό, ε, μάλλον χωρίς να επιβαρυνθεί ιδιαίτερο λογιστικός έλεγχος αυτών των κρατών. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ευχαριστώ. Δεν έχει ζητήσει κανένα άλλο το λόγο. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για όλες τις προτάσεις τους σε ό,τι αφορά τη μακροοικονομική βοήθεια, την ενίσχυση του προπολογισμού έγιναν κάποιες ε, προτάσεις, κάποιες παρατηρήσεις. Ξέρω ότι επιδέχεται βελτίωση και αυτό που έχω γράψει. Στο μεταξύ του ελεγκτικό συνέδριο έχει εκδώσει ειδική έκθεση. Ακριβώς για αυτό το θέμα, για τη δημοσιονομική ενίσχυση με προτάσεις για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά ήρθε αυτή η έκθεση μετά τη σύνταξη της δικής μου έκθεσης. και πώς ε, πηγαίνουν τα δημόσια κονδύλια στην απτυξιακή βοήθεια γιατί υπάρχουν και θέματα διαφθοράς. Μπαίνουν λοιπόν διάφορα ζητήματα, αλλά έχουμε και την πέμπτη την ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε αυτά. Ένα σχέδιο έκθεσης πάλι δικό μου, που είναι γνωμοδότηση για την πράσινη βίβλο που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μακροοικονομική βοήθεια τη δημοσιονομική ενίσχυση δηλαδή και υπάρχουν κάποια στοιχεία που δεν μπόρεσα να βάλω σε αυτή την έκθεση. Ξέρετε ότι έχω περιορισμό 2.000 ε, χαρακτήρες στην έκθεσή μου. Στη γνωμοδότηση μπορώ να το πω καλύτερα, αυτό που θα συζητήσουμε την Πέμπτη, και είναι γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας. Εν ανάγκη μπορούμε να το βάλουμε και στην έκθεση για την απαλλαγή με τροπολογίε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Είμαι πρόθυμο να δεχτώ όλε τι τροπολογίε, σα αν θέλετε να έχουμε και διμερεί επαφέ για να κοιτάξουμε πώ μπορούμε καλύτερα να διατυπώσουμε κάποια πράγματα. Και για τι ΜΚΟ κανένα πρόβλημα. Να γίνει με καλό τρόπο και... Έγιναν βέβαια κάποιε ερωτήσει, ειδικέ προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τον κύριο Έπινγκ, αλλά και από την κυρία Χόλμαγερ και από την κυρία Γκρέσλε για το καθεστώ του προσωπικού εκεί και να καταλάβουμε καλύτερα τι γίνεται με αυτού του υπαλλήλου. Και εγώ ρωτώ ως εισηγητή, θα μπορούσε να μα απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι τώρα, πριν τις 28 Μαρτίου και γραπτό, να μας δώσει μια καλύτερη εικόνα για να μπορούμε έτσι με τα λόγου γνώσεως και με ίσχυ τη συνείδησή μα να εγκρίνουμε ή να απορρίψουμε αυτές τις παραγράφους. Η να απορριψουμε αυτε τι παραγραφου η παρακαλώ. Πολύ σύντομα μερικά σχόλια σε αυτά που είπε η κυρία Χόλμαγερ καταρχήν για τους στόχους όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια είτε γεωγραφικά είτε κατατομής. Όντως αυτά αναφέρονται στην πράσινη βίβλο για τη νέα αναπτυξιακή πολιτική και στις, ε, στο νέο πολιετές ε, πλαίσιο. Όλα αυτά θα συζητηθούν. Βέβαια, ο επιμερισμός έχει ήδη γίνει για την τρέχουσα περίοδο δεν αναφέρθηκε μόνο η Βόρεια Αφρική. Γιατί εδώ δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό που συζητάμε για τη Βόρεια Αφρική. Πάντω η Επιτροπή θα συζητήσει την αντίδρασή τη για τη Βόρεια Αφρική. Δεν μπορώ να προδικάσω ποια θα είναι η έκβαση αυτής της συζήτησης. Πάντως η Επιτροπή μελετάει επισταμμένα επισταμένα τη νέα κατάσταση. Τώρα για τον εστιασμό σε νέες χώρε. Πολλέ από τι χώρες αυτές δεν είναι στη Βόρεια Αφρική και η Κομισιόν θέλει ε, να κοιτάμε και χώρες ε, για τις οποίες δεν πρέπει να είμαστε απόντε. Δεύτερο, προσλήψεις προσωπικού. Μιλάμε για προσωπικό στη κεντρική υπηρεσία, δεν είναι μόνιμη, συνδέονται με συγκεκριμένα ε, προγράμματα και maximum τρία χρόνια σύμβαση. Αυτό συμφωνεί απόλυτα με τις οδηγίες του Συμβουλίου σχετικά με τους, τα κονδύλια ιδίων πόρων για το προσωπικό. Τα ίδια κριτήρια εφαρμόζουν που έχει το Συμβούλιο. Για την κυρία Τσέσκοβα, σχόλιο για τα κοινωνικά. Ε, όντως, η, τα επιδόματα μητρότητας είναι ένα θέμα το οποίο καλύπτεται Γι' αυτό κινήσαμε μια ειδική διαδικασία προκειμένου να υπάρξουν κονδύλια επιπλέον για τις χώρες που θα έχουν εφερέγγια προγράμματα για το πάρα πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό μητρικής υγείας. Και κοιτάμε τα αποτελέσματα. Αυτό μας προσανατολίζει για να χρηματοδοτήσουμε χώρες που εφαρμόζουν τα μέτρα και όχι για κινήσεις προσανατολισμού να βάλουμε εκ των προτέρων 20% στην άκρη κονδύλια για, θέμα, για τέτοιου είδους στόχους που ενδεχομένως όμως να μην ε, εκπληρωθούν. Τέλος, για τον κύριο Έπινγκ για την, ε, ε, το ποσοστό απορροφητικότητας. Δεν έχουμε πρόβλημα εδώ. Μπορούμε να έχουν πλήρως δεσμευτεί τα κονδύλια και δίδονται στο 100%. Και το θέμα Βόρεια Αφρική δεν ισχύει στην περίπτωση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζοντας τον κύριο Έπινγκ, ξέρω ότι θα γράψει κανένα άρθρο τώρα ε, γνώμης και θα κυκλοφορήσει στις φλαμανδικές εφημερίδες. Ε, έχετε άλλες παρατηρήσεις? Όχι? Ωραία, τελειώνει και εδώ αυτό το θέμα. Την άλλη Δευτέρα το μεσημέρι στις 12 λίγη η προθεσμία για τις τροπολογίες και θα ψηφίσουμε στις 28 Μαρτίου. Έρχομαι στα διάφορα. Έχετε διάφορα? Όχι, κανείς. Ωραία. Η επόμενη συνεδρίαση την Πέμπτη στις 9 το πρωί. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ και τους διερμηνείς.